Iniziamo? Bene, cari colleghi, riprendiamo. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνουμε τι εργασίε μα. Έχουμε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο απογευματινό και α φροντίσουμε να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Πρώτο σημείο, προπολογισμό 2010, τμήμα τρίτον. Η συγγήτρια, η κυρία για Αγγλή για θέματα προϋπολογισμού. Γνωρίζουμε πως για την Γεωργία του 2010 θα αποτελέσει ένα έτος κρίσιμο σε ό,τι φορά την κατανομή κονδυλίων, αλλά τα περιθώρια θα είναι ιδιαίτερα στενά και τα περιθώρια αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια πολύ σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Επί του προπολογισμού έχουμε έχουν κατατεθεί 208 ε, τροπολογίες. 108 συγγνώμη. Η συγκήτριά μας, κυρία Γέγκλ, έχει παρουσιάσει την γνωμοδότησή της. Όλοι εργάστηκαν μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα και κατορθώσαμε να εργαστούμε αποτελεσματικά επί του θέματος, κάτι το οποίο δείχνει την βαθιά ανησυχία μας για το κατεπήγον ζήτημα και πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γεωργία, η οποία πλήττεται από την οικονομική κρίση και με κλάδους οι οποίοι διανύουν καιρούς πολύ σκληρούς. Εξετάσαμε σήμερα το πρωί το θέμα του γαλακτοκομικού τομέα. Έχουμε μια συζήτηση λοιπόν για την νομοδότηση και, για, και επί των τροπολογιών οι οποίε αύριο θα ψηφιστούν. Υπενθυμίσω πως η προθεσμία για την παρουσίαση ενεχόμενων τροποποιήσεων για το σχέδιο νομοδότησης έχει οριστεί η 9η Σεπτεμβρίου στις 12.00. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν επαναλαμβάνω το μεσημέρι στις 12. Και τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, κυρία Γέγκλη, για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες, αλλά και για το σχέδιο γνωμοδότησης. Υπενθυμίζω πως παρίστανται και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ο κύριο ε, Μπόκμαν, κυρία Μπόκμαν. Κυρία Γέγκλ, έχετε το λόγο. Äh, Ευχαριστώ. Äh, Ακούγεται δυστυχώς ένα βουητό στα ακουστικά μας και δεν ακούμε καλά την ομιλήτρια. Ναι, ναι, Σας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 το παραρελέ. Υπάρχει λοιπόν Α, ναι, υπάρχει, λοιπόν, λένε και άλλοι συνάδελφοι, παρεμβολή στα μικρόφωνα. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και θα διακόψουμε. Durchlesen und kritisch beachten. Im Gegensatz zu früheren Entwürfen, wo wir andere Probleme haben, hat dieser Entwurf natürlich den Hauptfokus auf den Milchsektor.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 Ευχαριστώ, λέτε τώρα μιλήτρια. Διορθώθηκε το πρόβλημα. Και έτσι λύθηκε και το τεχνικό πρόβλημα που δεν μας επέτρεπε να δουλέψουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, έχουμε τροπολογίες του... τις οποίες έχετε στο έγγραφό σας και θα ήθελα να ακούσω τις εκτιμήσεις σας κατά βάση Έχω ζητήσει να επαναφερθούν όλα τα ποσά όπου η Κομισιόν έκανε περικοπές. Δηλαδή, τροπολογίες τις οποίες μου δώσατε εμείς που αφορούν τη διαγραφή επιστροφών εξώσεων, ε, ε, εξαγωγών αποθήκευση και πριν, Όλες αυτές θα τις αρνηθώ, θα τις απορρίψω. Ακόμα και αν, και πιστεύω ότι οι επιστροφές εξαγωγών και η αποθήκευση δεν είναι τα κατάλληλα εργαλεία για το μέλλον. Η Κομισιόν μας έχει πει ότι τα μέσα αυτά, τα εργαλεία αυτά τα είναι πεπαλαιωμένα και θα πρέπει να τα διαγράψουμε. Μας έχουν πει ότι όλα αυτά δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, πρέπει να τα καταργήσουμε. Τώρα όμως φαίνεται ότι είναι η μόνη προσωρινή λύση την οποία μπορούμε να υιοθετήσουμε, δεδομένου ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για τους παραγωγούς και δι, οικονομικές λύσεις, χρηματοδοτικές λύσεις. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να μην, μην υιοθετήσουμε μια ριζική αλλαγή προς το συμφέρον, για το συμφέρον των παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το γαλακτοκομικό τομέα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 420 εκατομμύρια ευρώ έχω υπολογίσει μια νέα θέση για να υποστηρίξουμε το νέο οικονομικό περιβάλλον, το νέο οικονομικό περίγυρο Έχουμε βεβαίω και άλλα προγράμματα, αλλά από τα παλιά προγράμματα είχαν βγει τα 420 εκατομμύρια, αλλά εγώ τα ξανάλαβα. Άλλες τροπολογίες είναι τα οποροκυπευτικά. Πολλές φορές έχουμε κάνει αντίστοιχε ψηφοφορίες και υποστηρίζω αυτές τις τροπολογίες θετικές λοιπόν όπως και ε, την τροπολογία του κυρίου Σμιθ ε, για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ε, προβάτων. Για το γάλα είπα ότι έπρεπε να πω και για όσους ήρθαν τώρα θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Έχει εισαχθεί ως θέση στη συζήτηση μόνο επειδή πριν από δύο χρόνια έχουμε διαγράψει ορισμένα κονδύλια ε, που ανήκουν στην διοργάνωση της αγοράς και όταν διαγράφουμε κονδύλια που αφορούν την οργάνωση της αγοράς τότε αυτομάτως τα χρήματα αυτά ξαναπηγαίνουν στα κράτη-μέλη και εγώ ήθελα να προλάβω αυτή την κατάσταση έτσι ώστε τα ε, χρηματοδοτικά μέτρα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα να πρέπει να παραμείνουν στη διάθεσή μας το ρόλο που ορισμένα κονδύλια διαγράφονται στα πλαίσια της αντιοργάνωσης της αγοράς. Σήμερα το πρωί η κυρία Επίτροπος είπε ότι δεν συμφωνεί. Εγώ όμως είμαι πεπισμένη ότι αυτό το μέσο το χρειαζόμαστε, είναι μια πρόσθετη δυνατότητα των κρατών μελών να υποστηρίξουμε ε, τον γαλακτοκομικό τομέα. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα πιλωτικά τα οποία έχουμε υπερψηφίσει σε αυτή την Επιτροπή και θα πρέπει ε, να έχουμε και στη διάθεσή μας τα αντίστοιχα κονδύλια. Συνολικά εάν υπερψηφίσετε αυτά τα οποία προτείνονται, τότε θα υπερβούμε, θα υπερβούμε ε, γενικά ε, τις επιστώσεις. Οπότε θα πρέπει εμείς, να, κύριε Πρόεδρε, να αποφασίσουμε συνεχεία μέσα σε αυτή τη διαδικασία ψηφοφοριών ε, που μπορούμε να κόψουμε ώστε να τηρήσουμε τις προτεραιότητές μας. Εάν όλα υπερψηφιστούν, θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τις δυνατότητές μας, Διότι ο στόχος μας είναι γενικά να πετύχουμε την πλειοψηφία και στην Ολομέλεια και την, ε, την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Χέγγελ. Πραγματικά ήσταν σαφέστα ότι όλοι κατανοούμε την ε, σοβαρότητα του θέματος και την σημασία του. Ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά θα ολοκληρώσει η συγκήτριά μας. Ο κύριος Λουίς Σάντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ την κυρία Γέγκλ για την εργασία της. Ε, είμαστε συνηθισμένοι σε μια εξαιρετική εργασία, σε ολόκληρη τη θητεία της, ε, εργάστηκε εξαιρετικά. Συμφωνώ ως επιτοπλίστων με τις παρατηρήσεις σας, τις παρατηρήσεις της, Έχουμε και τον κύριο Φόλκο που είναι ο σκιώδης εισηγητής, ο οποίος δεν παρευρίσκεται δυστυχώς σήμερα αλλά είχε επαφέ με την κυρία Γέγκλ για να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ενημερώσω τους αδέλφου ότι η ομάδα των σοσιαλιστών προτίθεται να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό τροπολογιών, κυρίως αυτές που δίνουν μια απάντηση σε αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας θυμίζω και την πρωινή μας συζήτηση. Είμαστε επίσης διαθέσιμοι και προτιθέμαστε να ε, ε, εγκρίνουμε τις αλλαγές ε, για τις επιστροφές εξαγωγές για τα δημητριακά. Θυμάστε και την περσινή συζήτηση για το health check. Πάντως θα προσυπογράψουμε πάρα πολλές τροπολογίες αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες που είναι δημαγωγικές και θέτουν σε κίνδυνο τους συμβιβασμούς, ο οποίους έχουμε καταλήξει για να βρούμε μια διέξοδο για την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, οπωσδήποτε χρειάζεται αναθεώρηση, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τροπολογίε που συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση για κάποιου εκτροφεί των βοηδών Φερρυπίν. Πάντω θα έχουμε πολύ επικοδομητική στάση γιατί δεδομένων των δυσχερών συνθήκων ε, οφείλουμε να δώσουμε μία απάντηση ε, κυρίω για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που αντιμετωπίζει ο τομέα των γαλακτοκομικών και αυτή η απάντηση απάντηση πρέπει να δοθεί επίσης μέσα από τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Είναι απαραίτητο να στείλουμε κάποια μηνύματα. Επαντηλημένα ακούσαμε σήμερα αυτό το ζήτημα. Συμφωνούμε όλοι πως ε, οι προτάσεις της Κομισιόν δεν επαρκούν. Εργαζόμαστε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας μου ευχαριστώ την Ελίλη ε, για την εξαιρετική της εργασία και την ε, υποβολή πολύ θετικών προτάσεων. Βεβαίως ε, πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς όλοι. Ελπίζω αύριο στην ψηφοφορία να βρεθεί ένα τέτοιος καλός συμβιβασμός. Ήθελα μόνο να παρατηρήσω, επειδή και η κυρία Επίτροπος το ανέφερε, ε, ότι έχουμε περιορισμό κονδυλίου, περιορισμό πιστώσεων και επειδή υπάρχει αυτή η οικονομική πίεση θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε σε, αυτές, σε αυτή την επίγουσα και δύσκολη κατάσταση με τα υπάρχοντα μέσα Εάν όμως δει κανεί τα τεράστια ποσά τα οποία έχουν δοθεί από τις κυβερνήσεις για τη στήριξη των τραπεζών, τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί, δεν βλέπω γιατί δεν μπορούν να βρεθούν και κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης, ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και των παραγωγών. Κάνω λοιπόν μια έκκληση να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα κονδύλια, απαραίτητες πιστώσεις, ιδίως τώρα που υπάρχουν τόσο χαμηλές τιμές στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πρέπει πρέπει να ενισχύσουμε και την παραγωγή ε, τροφίμων και δι με, την πρώτη, με πρώτη ύλη το βούτυρο το, έτσι ώστε να μπορέσει το βούτυρο και τα προϊόντα βουτύρου να επανέλθουν και πάλι μέσα στη διαδικασία ε, της παραγωγής τροφίμων. Υπάρχουν ε, μεγάλες, ε, μεγάλα περιθώρια διάθεσης των προϊόντων αυτών. Βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές οι εξωτικέ χαμηλές τιμές στις γαλακτοποιικές μονάδες. Μην ξεχνάτε και το κόστος κιλού ανά βουτύρου. Και παλιά είχαμε τα τεράστια βουνά βουτύρου, θα θυμόσαστε, τα ιστορικά αυτά γεγονότα με τα 18 εκατομμύρια κιλά βουτύρου τα οποία είχαν συσσωρευτεί. Όλα αυτά τώρα έχουν εξαφωνιστεί αλλά δεν είναι δυνατόν να, να μην δώσουμε την ευκαιρία να ξαναχρησιμοποιείται αυτό το προϊόν έτσι ώστε να είναι ωφέλιμο για το, τους παραγωγούς και τις γαλακτοκομικές μονάδες τουλάχιστον να δώσουμε μια εναλλακτική λύση όσον αφορά την πρώτη ύλη και, την ενίσχυση του, των χαμηλών τιμών, όπως υποσχέθηκε η Επίτροπος. Ευχαριστούμε κύριε Γέγκερ για την εργασία σας, αλλά εμείς συνάγουμε διαφορετικά αποτελέσματα παρακολουθήσαμε τη συζήτηση το πρωί και συμφωνήσαμε σε ένα σημείο ότι σε ορισμένου τομεί θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική μα. Αλλά μα λείπουν οι λύσει. Τελείω. Εάν ακολουθήσουμε ε, την ε, κατεύθυνση τη σημερινή, δηλαδή ενίσχυση των εξαγωγικών πιστώσεων, τότε ακολουθούμε εσφαλμένο δρόμο. Πολύ βεβαίω μακροπρόθεσμα και κοντόφθαλμα να φτάσει αυτή η πολιτική, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι σωστή. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε και τις συνέπειες της ε, σημερινής συζήτησης, ε, το πρωί της πρωινής συζήτησης. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν την αγορά στα χέρια τους η παραγωγή Και γι' αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε με μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών τον τομέα. Δηλαδή θέλουμε τα χρήματα αυτά τα κονδύλια αυτά, τα οποία προβλέπονται για τις εξαγωγικές πιστώσεις, να πάνε στα χέρια των παραγωγών, δηλαδή να είναι χειροπιαστά λεφτά στα χέρια των παραγωγών που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να ενισχυθούν οι μονάδες τους. Πρόσφατα ακούσαμε τον εκπρόσωπο των γαλακτοκομικών ενώσεων της Νοτιού Αφρικής και μας είπε πώς έχει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Σε ορισμένες Βεβαίω υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση και στην Νότια Αφρική διότι υπάρχει αυτή η φθήνουσα πορεία των τιμών του γάλακτος και αυτό το, το, ε, το αρνητικό σπιράλι, ο έλικας αυτό, ο οποίο τίνει προ τα κάτω, προ τι χαμηλότερε τιμέ. Γι' αυτό πιστεύω ότι και επαναλαμβάνω, αντί για ενίσχυση των εξωτερικών πιστώσεων, τα χρήματα αυτά να πάνε στα χέρια των παραγωγών για την ενίσχυση του γαλακτοκομικού τομέα και των τιμών των προϊόντων. Ευχαριστώ. Μόρουεϊ, έχεις τη στο λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι δεν ε, βλέπω να έχει προωθηθεί το ιδέα της ε, κοινωνικής πολλαπλής συμμόρφωσης ε, που είχα προτείνει το πρωί. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε κάποια ευθύνη και να μπορέσουμε με τρόπο αυτό να επιλύσουμε την, το πρόβλημα και να διατηρήσουμε τις θέσεις ε, απασχόλησης ε, στην γεωργία. Διότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η βάση της προτασιός μου ήταν το άρθρο 39 της Συνθήκης Ρώμης, το οποίο αναφέρει πως η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να έχει ως στόχο αποσιοποιητικά διάφορα και την βέλτιστη χρησιμοποίηση των ε, παραγόντων παραγωγής ε, και δι της ε, εργασίας. Βλέπετε λοιπόν ότι η δική της Ρώμης μιλάει και για την εργασία και όχι μόνο για το κέρδος. Εγώ θα ήθελα να προτείνω λοιπόν να διατηρηθεί το 10% των επιδοτήσεων του γαλακτοκομικού τομέα και των και του σε νέα ενίσχυση, και να πάρουμε το 5% προκειμένου να μπορέσουμε να εισαγάγουμε αυτήν την νέα επιδότηση η οποία θα χορηγείται στους γεωργούς οι οποίοι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν θέσει εργασία. Τι θα σημαίνει αυτό για το τη γεωργία, ότι υπάρχει μια μικρή εκμετάλλευση όπου εργάζεται ο σύζυγος. μέσω αυτής της επιδοτήσεως θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια δεύτερη θέση εργασία είτε για τη σύζυγό του και χαίρομαι που αυτή η πρόταση είναι τόσο από από από τους συναδέλφους εδώ γύρω και θα μπορούσαν λοιπόν να παράγουν κάποια προϊόντα όπως ε, τυριά αυτές οι εκμεταλλεύσεις. Εδώ έχω δύο σελίδες ε, που αιτιολογούν την ε, τροπολογία μου όπου καταδεικνύω πως ε, θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια πρόταση υπέρ των γεωργών στην Ευρώπη και να δώσουμε μια μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Και έτσι θα μπορούσαν να παροτριθούν οι γεωργοί στο να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιδοτήσεις για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις οικογένειάς τους, στις κοινωνίες τους κλπ. Θα ήθελα να ακούσω κάτι λοιπόν από την εισηγήτρια περί αυτού. Ποια λοιπόν με λίγα λόγια θα είναι η αντίδρασή της σε αυτή μου την πρόταση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι παρεμβαίνοντες, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα στην κυρία Μπότσμαντ θα ακολουθήσει η συγγήτρια. Παρακαλώ, κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σχόλια στο σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την πρόταση περί αποκατάστασης του προσχεδίου προϋπολογισμού που κάνει η συγγήτρια προτείνει να καταργήσει δηλαδή τις περικοπές του Συμβουλίου. Επίσης, στο σχέδιο καλωσορίζουμε την αναφορά στην τροποποιητική επιστολή. Διάφορες τροπολογίες που υποβάλλατε εσείς θα εξεταστούν από την Επιτροπή μέσα στην ε, τροποποιητική επιστολή που θα έχουμε ετοιμάσει μέχρι τον Οκτώβρη, όπου θα επανεξετάζουμε την τωρινή κατάσταση στην αγορά συμπεριλαμβανομένου και το τομέα των γαλακτοκομικών και οποιαδήποτε άλλα ε, συναφή ζητήματα. Θα δούμε ποια κομμάτια της πρότασής μας δηλαδή πρέπει να τροποποιήσουμε και αν ε, χρειάζονται περαιτέρω δαπάνες. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφέρω το πόσο σημαντικό είναι για τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και για την γενικότερη ανάπτυξη του τομέα να Έχουμε την 050145, τη νέα γραμμή του προπολογισμού, η οποία θα επανενταχθεί στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν γίνουν οι περικοπέ από το Συμβούλιο σε αυτέ τι γραμμέ, ε, δεν δύνατη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαταστήσει τη 0514 γιατί σε αυτήν βασιζόμαστε για τις αξιολογίες και τις μελέτες που κάνουμε που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναθεώρηση και του προϋπολογισμού και γι' αυτό καλωσορίζουμε αυτή την πρόταση της εισηγήτριας. Για το γαλακτοκομικό τομέα τώρα ε, το πρωί συζητήθηκε το θέμα και μίλησαν άλλοι εκπρόσωποι, συνάδελφοί μου, δεν έχω να προσθέσω εγώ τίποτα. Ε, για το σύστημα για την διανομή φρούτων ε, στα σχολεία. Το ποσό που προβλέπεται για το 2009-10, τη σχολική χρονιά, είναι 9 εκατομμύρια. Αυτό προβλεπόταν στην αρχική πρόταση, αλλά υπάρχουν και κάποιε τεχνικέ πτυχέ στο προπολογισμό. Αυτό σημαίνει το τελευταίο τρίτο θα ε, καταβληθεί το 2011. Γιατί ε, τελικά τις, ε, θα υποβληθούν οι τελικέ αιτήσει για αποζημίωση από τα σχολεία στο τέλο του σχολικού έτου και μέχρι να επεξεργαστούμε εμεί τι αιτήσει θα φτάσει το 2011, γιατί πρέπει να γίνουν και έλεγχοι από πλευρά μα. Ε, προβλέπεται λοιπόν αυτό το αρχικό ποσό, τα 90 εκατομμύρια, αλλά θα πληρωθούν ουσιαστικά κατά αυτό το σχολικό έτος μόνο τα 60 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει κατόφλι για αυτό το σύστημα, για τα σχολεία, δηλαδή ε, μπορούν να δαπανηθούν κάποια κονδύλια από τα κράτη-μέλη ως υποχρεωτικές δαπάνες και να σας πω ότι φέτος παραφερειπίνε τα κράτη-μέλη ε, δαπάνησαν περισσότερες πιστώσεις από αυτές που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού για το σύστημα, για τα σχολεία. Τώρα, κάποια γενικά σχόλια για τις τροπολογίες. Βλέπω διάφορες τροπολογίες που ευθυγραμμίζονται με τα συμπεφωνημένα στα πλαίσια του health check. Ε, ας πάρω ένα παράδειγμα. Ε, για το λινάρι και την κάναβη ε, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις από το 2010. Οπότε ε, ε, συνάγουμε ότι έχουν συμφωνηθεί ήδη αυτές οι προτάσεις στα πλαίσια του health check. Τώρα για τα περιθώρια. Λέτε εσείς ότι έχουμε ένα σε περιθώριο. Ναι, αλλά αυτό είναι για το συνολικό, για το κεφάλαιο 2. Ε, για τον πρώτο πυλώνα έχουμε μόνο 1 δις περιθώριο, δηλαδή 100 εκατομμύρια λιγότερο. ένα δις. Αυτά για τον πυλώνα 1 και εκεί θα εφαρμοστεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Αν δείτε ποσά από την Επιτροπή που μιλάνε για 1,1 δι σε περιθώριο, ε, ε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το υποκατόφλι για τον ε, πρώτο πυλόν. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω, κατάλαβα δεν έχουμε να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστούμε την κυρία Μπόρσμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γέγκλ να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση έτσι ώστε αύριο θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τους συναδέλφους που παρενέβησαν και την εκπρόσωπο της Κομισιόν ευχαριστώ επίσης. όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν είχαν ένα στόχο βασικά. Τους παραγωγούς. Τους παραγωγούς και τη στήριξή τους. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το ερώτημα είναι πώς θα εκπληρώσουμε αυτό το στόχο. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις σας, ε, τα αιτήματά σας. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αλλά βασικά στη διαδικασία προϋπολογισμού δεν μπορούμε να εισάγουμε μια νέα αγροτική πολιτική, μια νέα γραμμή αλλά πρέπει να τα βγάλουμε πέρα με αυτά που έχουμε. Ε, είπε η Επίτροπος ότι έγινε το, το, το τσεκάρισμα της υγείας, ο έλεγχος υγείας, έγινε επίσης ε, η μεταρρύθμιση ε, της ΚΑΠ ε, και εγώ βεβαίως έχω πολλά ερωτήματα στο μυαλό μου με την σημερινή κατάσταση αλλά έχουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και σε αυτά πρέπει να βασιστούμε. Ο προϋπολογισμός του 2010 είναι βράχη πρόθεσμος προϋπολογισμός. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη συζήτηση για το μέλλον, μακροπρόθεσμα δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες βάσεις. Αυτό ισχύει και για σας κυρία Μόβλη. Εξέτασα με προσοχή τις ε, τροπολογίες σας και με έβαλαν σε πολλές σκέψεις. Δεν έχουμε μια νομική βάση, ένα νομικό υπόβαθρο να υιοθετήσουμε κάτι τέτοιο. Και μέσω του προϋπολογισμού να κάνουμε μια τέτοια μεταρρύθμιση στην αγροτική πολιτική δεν νομίζω να γίνεται. Βεβαίως ε, η πρότασή σας ε, έχει αξιόλογα στοιχεία αλλά για αυτό τον κατάλογο τροπολογιών που έχω να ψηφίσουμε αύριο, σας παρακαλώ να κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε άλλες τροπολογίες. Έχει κλείσει ο κατάλογος. Ε, επίσης, το ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε 10% από τις ενισχύσεις ή από τις ε, αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις τους ε, τώρα είναι κατανοητό για να καλύψουμε, ε, ε, εάν κάναμε αυτές τις περικοπές, θα έπρεπε να πούμε ταυτόχρονα στους, γεωργούς, στους παραγωγούς ότι κάτι άλλο θα βρούμε να σας αποζημιώσουμε, που δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και ευχαριστώ την Κομισιόν. Θα πρέπει μαζί όλοι να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τα πλαίσια, τα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού και των δαπανών πρέπει επίσης να πιέσουμε και σε εθνικό επίπεδο τους συναδέλφους μας, τα Υπουργεία, τους αρμόδιους, να διαθέσουν τα κονδύλια αυτά που, που χρειάζεται η Γεωργία. Για τα φρούτα και το γάλα, ε, τονίζω και πάλι ότι τα δύο προγράμματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Σήμερα το πρωί ζητήθηκε η πρόθεση του γάλακτος ως προϊόν και ίσως να προσφέρετε εδώ γάλα και εδώ στην Ολομέλεια και στο Στρασβούργο. Εντάξει, καλό είναι σε εμά να διατίθεται το προϊόν, αλλά περισσότερο πιστεύω και στα παιδιά, στα σχολεία χρειάζεται η ενίσχυση της ζήτησης για φρούτα, για γάλα και πιστεύω ότι τα κράτη θα χρησιμοποιήσουν, τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν σωστά τα κονδύλια αυτά που τους δίνουμε για την προώθηση των προϊόντων αυτών, φρούτων και γάλακτος. Ευχαριστώ. Ωραία. Στο σημείο αυτό νομίζω πως ολοκλώσαμε το σημείο 5 της μεσαίας διατάξεως και αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε υπενθυμίζοντας πως αύριο πρόκειται να ε, περάσουμε στις ψηφοφορίες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες ε, προκειμένου να εγκρίνουμε τις τροπολογίες. Grazie. Ε, mi faceva segnalare di μου υπενθύμησαν πως θα πρέπει με τη σειρά μου να σας υπενθυμίσω δεδομένου του ότι αύριο πρόκειται να ψηφίσουμε να φέρετε όλοι τις ε, κάρτες σας ε, έτσι ώστε να είστε σε θέση να ψηφίσετε. Μην ξεχάσετε λοιπόν, μην λησμονήσετε τις ε, κάρτες. Περνάμε στο σημείο 6. Πρόκειται για την παρουσίαση μιας μελέτης για τον ΠΟΕ, μια ανταλλαγή απόψεων. Θα μας γίνει μια σύντομη παρουσίαση. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Όλιβερ Πρόστο και τον κύριο Μαξίμ Προυντέν που θα μας μιλήσουν για τις διαπροντεύσεις στο πλαίσιο της ΠΟΕ μετά από την αποτυχία, τη χρεοκοπία των συζητήσεων 2008. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό μα το οποίο θύμισε και η Επίτροπο σήμερα το πρωί, θα διαβάσατε κι εσείς ε, την ε, επίσημη διακήρυξη των ε, και δέσμευση των ε, υπευθύνων να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία. Είναι ένα ζήτημα ζωτική σημασία. Ε, θα πρέπει να ακούσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης και να περάσουμε αργότερα σε μια συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Πρόστ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέλη του Κοινοβουλίου. Κοινοβουλίου. Το όνομά μου είναι Ολιβία Πρόστ και μας ζητήθηκε να προετοιμάσουμε μία μελέτη για τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕΣ, τις αγροτικές, γεωργικές διαπραγματεύσεις και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μπορούμε να ε, παρουσιάσουμε αυτήν την έκθεση στη Νέα Επιτροπή Γεωργίας. Είναι λίγο δύσκολο στα 20 λεπτά αλλά θα προσπαθήσω. Μία σημαντική πρόκληση λοιπόν καταρχάς είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν διαφορετικά αγροτικά μοντέλα και έτσι έχουμε αντιφατικές ε, ε, πτυχές, αντιφατικές ε, ιδέες και πραγματικότητες. Από τη μία πλευρά έχουμε την απελευθέρωση, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και την επιθυμία διατήρησης ορισμένων γεωργικών πολιτικών και μπορούμε να πούμε ότι σήμερα τα μέλη έχουν πλέον δεχτεί την μέγιστο, το μέγιστο βαθμό απελευθέρωσης, ο οποίος είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτός. Βεβαίως οι διαπραγματεύσεις αυτές αφορούν έναν, ε, ένα αναπτυξιακό πλαίσιο. Είναι ένας γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο την ανάπτυξη και θα οδηγήσει σε ασύμετρες ε, παραχωρήσεις. Αυτή η ασυμμετρία ε, θα δημιουργήσει μια πιο δύσκολη κατάσταση. Εμείς επιθυμούμε να ακολουθήσουμε μια ενιαία κατεύθυνση και να επιτύχουμε μία ισορροπία μεταξύ διαφορετικών και ασχέτων ε, θεμάτων, γεωργικών και μη γεωργικών υπηρεσιών και, και εκτός υπηρεσιών. Ε, ένας μεγάλος αριθμός ε, διαπραγματευτών ασχολείται με αυτά τα θέματα και γίνονται διαπραγματεύσεις και έντονες συζητήσεις με τις αναπτυσσόμενες και νέες βιομηχανικές χώρες, ε, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Κίνα. Το, οι επιπτώσεις των παραχωρήσεων έχουν άμεση σχέση με την περιπλοκότητα των λύσεων που προτείνονται. Ε, αν θέλετε μία μείωση των δασμών, θα πρέπει παράπλευρα να εφαρμόσουμε μία ε, ελαστικότητα σε άλλες πολιτικές και αυτά όλα έχουν διαφορετικές επιπτώσεις. Είναι και δύσκολη εκτίμηση των επιπτώσεων. Αυτές λοιπόν είναι οι προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά ε, πρέπει να πω ότι ζητούμε σήμερα ένα πακέτο ε, το οποίο στην ορολογία του ΠΟΕ λέγεται draft modalities. Έτσι λέγεται αυτό το πακέτο. Και θα σας εξηγήσω τι εννοούμε με αυτόν τον όρο, modalities. Το πακέτο αυτό τα περιλαμβάνει καταρχάς μέτρα για την χώρια ενίσχυση. Δηλαδή, να ενισχυθούν ε, οι πειθαρχίε ε, για την ενίσχυση των ε, μέτρων εξομάλυνσης των στρεβλωτικών πτυχών του εμπορίου. Η ρήτρα δεσπόζουσας θέσης θα μειωθεί κατά 50% και προτείνουμε και ένα άλλο, μια άλλη όροφη η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί σε περίπτωση στρεβλωτικών μέτρων όπως μίνιμουμ ε, ποσοστά, το μπλε κουτί, το πράσινο κουτί και διάφορα άλλα τέτοια μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν την οροφή ε, ορισμένων προϊόντων. Όσον αφορά το πράσινο κουτί, οι ενισχύσεις εδώ θα δίνονται με πολύ αυστηρότερα κριτήρια έτσι ώστε να έχουν ελάχιστες στρεβλωτικές επιπτώσεις δεν θα υπάρχουν όρια στον προϋπολογισμό μεν, αλλά νέες πειθαρχίες θα εισαχθούν πολύ σημαντικά, ιδίως για τις αποσυνδεδεμένες πληρωμές. Εκτός αυτού θα υπάρχουν και πολλές, ε, ε, πολλά ευέλικτα μέτρα σε εισαγωγικά που θα ε, παραχωρηθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες παράταση περιόδων, μείωση ενισχύσεων για το βαμβάκι και επίσης άλλα μέτρα μέσα στο πλαίσιο, στα πλαίσια του Black μπλε κουτιού, blue box, αυτή η ενίσχυση λοιπόν μέσα στο, του Blue Box θα οριοθετηθεί, θα έχει ένα συγκεκριμένο, ε, μια συγκεκριμένη οροφή και με τις συζητήσεις που γίνονται με τις Αμερικανούς εταίρους θα εξετάσουμε ε, τη δυνατότητα ε, απόσυρσης ε, του καταλόγου προϊόντων, του περιορισμού δηλαδή της εφαρμογής του Blue Box σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο προϊόντων. Έτσι το ζήτησαν οι Αμερικανοί. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση στην αγορά, εδώ προβλέπονται περισσότερες, περισσότερα πειθαρχικά μέτρα, αλλά και μείωση των προσκομμάτων πρόσβασης ποσοστώσεις δασμών, κλιμακωτή διάστρωση των δασμών και ένας κατάλογος ευαίσθητων προϊόντων έτσι ώστε να μπορούσαν οι χώρες αυτές να ε, ελέγχουν ε, την ε, κατάσταση που επικροτεί στα σύνορά τους μαζί με την, με ταυτόχρονη επέκταση των ποσοστώσεων δασμών. Special οι δασμοί τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, ε, μέσα στα πλαίσια της Ιρουάης έχουν χρησιμοποιηθεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα ε, ενδέχεται βεβαίως ε, για την πρόσβαση στην αγορά να εισάγουμε ορισμένα ειδικά προστατευτικά μέτρα για αναπτυσσόμενες χώρες που θα καλύπτουν ειδικά προϊόντα, ευαίσθητα, ειδικά, ειδικές ρήτρες ασφαλείας, ε, ειδικοί μηχανισμοί ε, ασφαλείας, τα Special Safeguard Mechanisms και άλλους κανόνες, όλα αυτά για την ειδική προστασία αναπτυσσομένων χωρών. Στην, ε, στον ανταγωνισμό εξαγωγών, στον εξαγωγικό ανταγωνισμό, εδώ προβλέπουμε την βασμιαία μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων μέχρι το 2013. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα των εξωτερικών χωρών αλλά και πολλών αντισωμένων χωρών και ταυτόχρονα θέλουμε να ενισχύσουμε την τους, ε, την πειθαρχία στους τομείς, την σωστή διοργάνωση δηλαδή, ε, με άλλα κίνητρα εξαγωγικά, όπως ε, προγράμματα εξαγωγικών πιστώσεων, κρατικές εξαγωγικές διευκολύνσεις και ενίσχυση αγοράς τροφίμων. Τον ε, Ιούλιο του 2008 ο, είχε, ο Πασκάλ Αμή πριν από τον Ιούλιο του 2008 είχε προτείνει ε, ένα πακέτο μέτρων στον αγροτικό τομέα που περιλάμβανε όμως και, όχι, και μη αγροτικά θέματα τα οποία αναπερίφθηκε τον Ιούλιο του 2008. Η ιδέα ήταν να μειώσουμε τις τρευλώσεις ε, του ε, τομέα, να μειώσουμε τους δασμούς και να δεχθούν τα μέλη το προτινόμενο αυτό πακέτο. Μείωση δασμών, απελευθέρωση ειδικών τομέων, ε, ρήτρα κατά της συγκέντρωσης του anti-concentration. Όμως απερίφθηκε, όπως είπαμε, αυτό το πακέτο λαμή και έτσι τελικά παρόλα αυτά έγινε σημαντική πρόοδος σε αρκετά θέματα ε, αλλά εκφράστηκαν και πολύ μεγάλες επιφυλάξεις, ειδικά από την Αμερικανική πλευρά, ότι η υπερβολική ευελιξία θα εξουδετερώσει ε, τις, ε, τα μέτρα απελευθέρωσης. Εάν προσπαθώντας τώρα να εκτιμήσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της ΚΑΠ, μπορούμε να πούμε τα εξής. Για τις επιδοτήσεις συνολικά θα πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια με τα μέτρα του, της Ντόχα ε, και με τη σημερινή ΚΑΠ τα οποία να στοχεύουν λιγότερο στις τιμές και στην διακύμανση των εισοδημάτων από ότι η αμερικανική πολιτική. Υπάρχουν δυνατότητες να δοθούν σημαντικές ενισχύσεις ε, σε περιπτώσεις τρέβλωσης του ανταγωνισμού, ε, του εμπορικού ανταγωνισμού αλλά και ε, των εισοδημάτων και πιστεύουμε ότι τα επίπεδα ενίσχυσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υπάρχοντα όρια που είναι 22 δις για την ε, μη εμπορική ενίσχυση ε, και 40 δις για το πράσινο κουτί, για τις ε, γεωργικές ενισχύσεις. Ε, τώρα, για την πρόσβαση στην αγορά. Σημαντικέ μειώσει του δασμού σε 60% κατά μέσο όρο θα αυξήσουν ασφαλώς την εξωτερική έκθεση στον ανταγωνισμό και στην ε, διακύμαση των τιμών. Ταυτόχρονα όμως τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ειδικά μέτρα προστασίας για τα ευαίσθητα προϊόντα για τα οποία όπως σας είπα ήδη έχουμε ζητήσει επέκταση του χρόνου των προθεσμιών ιδίως για τα προκυπευτικά για τον, για τον εξαγωγικό ανταγωνισμό ε, μείωση των, ε, εξαγωγικών, επιστροφών μέχρι το 2013 σύμφωνα με την αναθεώρηση της ΚΑΠ και επίσης ανάγκη αμοιβαίων μέτρων υπό την μορφή εξαγωγικών ε, κινήτρων, παροχής εξαγωγικών κινήτρων. Τώρα, η αξιολόγηση της αμερικανικής έναντι, ε, θέσης έναντι της αμερικανικής γεωργικής πολιτικής. Καταρχάς, εγχώρια ενίσχυση. Εδώ η, τα προτινόμενα μέτρα της Ντόχα δεσμεύουν σημαντικά τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί ένα μεγάλο μέρος των άμεσων πληρωμών στην Αμερική δίνεται ακόμα μέσα στο... Ε, μέσα στο μπλε και κίτρινο κουτί ενώ οι περισσότερες ε, ε, ε, στηρίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα του πράσινου κουτιού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία ρήτρα de minimis για την διαθεσιμότητα των ενισχύσεων και αυτή η ρήτρα, το, όριο αυτό θα μειωθεί. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα χρειαστεί να εφαρμόσουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για τον ανταγωνισμό, ε, τον εξαγωγικό. Θα, δω, θα προτείνουμε, ε, γίνονται διαβουλεύσεις για τις επιστροφές εξαγωγών και για την επισητιστική βοήθεια όπου χρειάζεται αναθεώρηση. Για την πρόσβαση στην αγορά το πιο σημαντικό μέτρο δηλαδή για τους Αμερικανούς είναι ότι ε, χρειάζεται μια φιλόδοξη φόρμουλα για τη μείωση των δασμών ε, υπάρχουν βέβαια αμερικανικές επιφυλάξεις όσον αφορά το εύρο των ε, ευέλικτων μέτρων ευελιξίας που δίνουμε στι αναπτυσσόμενες χώρες και τι επιπτώσεις έχουν στην πρόσβαση στην αγορά. Τώρα, οι συνολικέ επιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, αρνητικέ επιπτώσει δεδομένου ότι αυξάνονται οι εισαγωγέ. Αύξηση ε, εισαγωγών ίσον αρνητικέ επιπτώσει. Δεύτερον, ίσως θετικές επιπτώσεις στο θεμητό ανταγωνισμό ως αποτέλεσμα των πιο ισχυρών ε, πειθαρχικών μέτρων που θα εφαρμιστούν ε, και επίσης των εξαγωγικών κινήτων που θα δοθούν. Ενδεχομένως καλύτερη πρόσβαση στην αγορά ε, τρίτων χωρών και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με, τις, με τα ευέλικτα μέτρα που θα δοθούν σε αυτές τις χώρες. Οι δυνατότητες της ΚΑΠ θα πρέπει να ε, μη στρεβλώνουν ε, τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα και τέταρτον η επίπτωση και πέμπτον η επίπτωση των οικονομικών ε, προβλέψεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τους τομείς του ΠΟΕ. Πριν κλείσω θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την ερήτρα ειρήνης. Ε, επειδή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις, ε, μπορεί να αυξηθούν οι διαφορές στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αλλά ακόμη και αν τελικά ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις, κάποια μέλη του ΠΟΕ μπορεί να έχουν συμφέρον να αποφύγουν τις δικαστικές διαφορές, όπως ε, για τη συμφωνία για τις ενισχύσεις των εξαγωγών, των εγχωρίων εξαγωγών. Παραδείγματος χάρη στο ΠΡΑΣ, υπάρχουν μέτρα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ε, ε, ε, συνεπάγονται επιβλαβή μέτρα για την εγχώρια οικονομία. Τέτοιου είδους διατάξεις μπορούν να εξεταστούν στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η ΕΠΑ μπορεί να έχουν συμφέρον να ζητήσουν υιοθέτηση νέα ρήτρα ειρήνη που θα αναστάλει προσωρινά την εφαρμογή τη συμφωνία για τι ενισχύσει εν ώψη και των τελευταίων εξελίξεων στην ομολογία του ΠΟΕ στην περίπτωση, στην υπόθεση για το βαμβάκι ή για τη ζάχαρη. Ε, εξαρτάται από την ερμηνεία του σώματος για τις εφέσεις. Οι παράμετροι όμως δεν έχουν προσδιοριστεί για μια πιθανή συμφωνία. Ε, ποιες είναι οι προοπτικές. Ε, ε, μία συμφωνία για το τωρινό πακέτο, όπως σας είπα, για βασικά ζητήματα όπως τα ευπαθή προϊόντα ειδικέ ρήτρε διασφάλιση για τι αναπτυσσόμενε χώρε, ε, για διεύρυνση των ευέλικτων διατάξεων κτλ. και κάποια άλλα ζητήματα που δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η ρήτρα ειρήνη για τι ε, ΗΠΑ ε, και οι G20, οι G33 εργάζονται Εσχάτως, για αυτά τα ζητήματα και στα πλαίσια του ΠΟΕ συνεχίζονται οι εργασίες. Θα δούμε, αναμένουμε τις εξελίξεις. Ε, άλλη πιθανή έκβαση είναι το μπλοκάρισμα η αποτελμάτωση της κατάστασης δηλαδή μπορεί να καταλήξουμε σε μίνι πακέτα για το αναπτυξιακό θέμα αλλά αυτό δεν είναι πολύ πιθανό. Μπορεί επίσης να ε, συζητηθεί ε, να γίνει ένας, μια από κοινού συζήτηση πολυμερών και διμερών ε, ζητημάτων σχετικά με τις ευέλικτες διατάξεις εξαρτάται από τα συμφέροντα κάποιων κρατών μελών ή Ε, μπορεί να ε, δούμε αύξηση των ε, δικαστικών διαφορών για μη δασμολογικούς φραγμούς, για εγχώριες ενισχύσεις ή και μπορεί να αναπτυχθούν νέες διμερείς ή περιφερειακές προσεγγίσεις ή μπορεί να σημειωθεί αύξηση του φαινομένου και των δύο αυτών προσεγγίσεων εκ τι, ποια είναι η πιθανή προσαρμογή τώρα στα πλαίσια του ΠΟΕ της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα είναι απίθανο να καρκινοβατήσουμε, να επιστρέψουμε στο παλιό ε, σύστημά μας, ε, δηλαδή παρεμβατικό σύστημα, αύξηση των ενισχύσεων ε, προς για τις εξαγωγές, ε, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέε ενιαίε ενισχύσεις με μια καλύτερη κατανομή των ενισχύσεων ε, στις εκμεταλλεύσεις σαν γεωγραφική ζώνη και αν δεν αρκέσει αυτό μπορεί να παραταθούν τα τωρινά συστήματα συγχρηματοδότησης και ταμείων αλληλεγγύης, αλλά μπορεί να υπάρχει και παρέμβαση σε ευαίσθητους τομείς, όπως ε, και σχετικά με τα κίνητρα των, του ΠΟΕ, που κρίνονται συμβατά με τις διατάξεις του ΠΟΕ. Επίσης, για να προστατευτούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πιο παραδοσιακά εργαλεία, για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των γεωργών ε, μέσα από ενισχυμένες ιδιωτικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και ενίσχυση των σχέσεων ε, και του συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Πρόστο για αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη. ότι εμείς έχουμε διανύμει αντίγραφο σε όλους τους συναδέλφους. Θεωρώ πως ε, είναι σημαντικό το ότι εστιάσατε το πρόβλημα και διότι το ζήτημα αυτό θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στι προσεχείς εβδομάδες και μήνες ε, και στο πλαίσιο του νέου ρόλου που πρόκειται να αποκτήσει το Ευρωκοινοβούλιο μετά από την Δευτέρα Οκτωβρίου εάν όλα πάνε καλά. Να δώσω το λόγο τώρα στους πρώτο Πρώτος ε, έχει το λόγο ο κύριος Λάτενφέρντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω στον Γκρικά, αφού μπορώ. Μία, η φωνή της μέσης Ευρώπης. Με την γλώσσα μου, λοιπόν. Αν λάβουμε υπόψη τι κανονισμούς γλωσσικούς κανονισμούς έχει εισάγει γάγει η Σλοβακία, καλύτερα να μιλήσω ουγγρικά, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η βάση της, ε, του γύρου της Ντόχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να συζητηθούν τρία σημαντικοί, τρεις σημαντικοί τομείς και ε, ο τομέας της γεωργίας ε, απαιτεί συνεχώς παραχωρήσεις και υποχωρήσεις ε, διαφορετικές από τους τομείς της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των άλλων δύο τομέων και του αγροτικού. Και πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα στον αγροτικό τομέα δεν είναι αποδεκτά πλέον. Έχουμε τώρα μια εντελώς καινούργια οικονομική κατάσταση και γι' αυτό το θέμα αυτό έχει προσλάβει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε η οικονομικές, ε, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ούτε ε, οι εξαγωγικές διαδικασίες μπορούν να επιτρέψουν ε, ή η, ενίσχυση της βιομηχανίας μπορεί να επιτρέψει την, τον παραγωνισμό του αγροτικού τομέα. Γι' αυτό με αυτή την κρίση που υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην προσέξουμε τις ε, λεπτομέρειες, τα μικρά γράμματα μόνο, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο. Πώς θα προχωρήσουμε μετά το γύρο της Δόχα, πώς θα προχωρήσουμε πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ακολουθήσει έναν εσφαλμένο δρόμο μέχρι τώρα, πρέπει από εδώ και μπρος να ακολουθήσουμε τη σωστή οδό. Ωραία. Η κυρία Εραντ Γκαρσία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως το επίκεντρο της συζήτηση θα πρέπει να αποτελέσει η τελευταία πρόταση που μας είπε ο εμπειρογνώμων, δηλαδή καλύτερη προστασία του ευρωπαϊκού συμφέροντος και οι ανησυχίες μας τόσο για το περιβάλλον μέσω μια ε, καλής εταιρική σχέση ιδιωτικού δημόσιου τομέα, μια σύμπραξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι κράτησε λάθος ε, στάση από την αρχή των διαπραγματεύσεων. πάντω η γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν ένα ζήτημα συνδιαλλαγή και δεν ε, μας δίναμε μέσα ενδιαφέρει διόλου το αποτέλεσμα. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πως δεν είναι των ίδιας απόψεως και δεν φροντίζει να σεβαστεί τα δικαιώματα. Και ως αποτέλεσμα ήταν ε, τα ευαίσθητα προϊόντα να μην αναγνωριστούν και να βλέπουμε συνεχώς παραβιάσεις των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας λέει για ποιο λόγο με... δεν γίνεται συστηματικός έλεγχος των προϊόντων τρίτων χωρών και υπάρχουν και κάτι άλλα θέματα που μα ανησυχούν ιδιαίτερα μετά από όσα ακούσαμε. Πάντως φαίνεται ότι οι πληρωμές των, πολιτιών καταλήγουν στο μπλε κουτί και άρα θα νομοποιηθούν. Η κοινή αγροτική πολιτική μας έχει όλο και λιγότερα χρήματα για να βοηθήσει τους γεωργούς και εμείς α, κάνουμε με ένα είδος αυτοπερικοπών. Από ό,τι γνωρίζω η Ευρώπη πάντα ε, σεβάστηκε τις ε, δεσμεύσεις κατά 120%. Τώρα πώς θα αρχίσουμε να αξιολογούμε αν οι ε, αναδυόμενες χώρες έχουν ήδη αναδυθεί, αναδυθεί όπως η Κίνα, η Βραζιλία, οι, Αφρικανικές. Δεν μπορούμε να θεωρούμε συνεχώς ως αναδυόμενες, ορισμένες έχουν ήδη αναδυθεί και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να λιχάνουν αυτή τη αντιμετώπιση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη καταστεί ισχυρέ δυνάμει. Τώρα και ποια είναι η θέση των ΗΠΑ, διότι οι αντικυκλικέ ενισχύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και εμεί βρισκόμαστε πάντα Ένοχή και δαχτυλοδεικτούμενοι. Θα ήθελα επίση να γνωρίζω τι έγινε με τις προηγούμενες συμφωνίες, αν έχουν τηρηθεί και με ποια μορφή. Ποια θέση λοιπόν πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσεχείς διαπραγματεύσεις προκειμένου να τηρηθούν οι συμφωνίες. Και μιλάμε τώρα για προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τρίτων πρωινών τρίτων χωρών, τη φορά την χνηλασιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν αυτέ τι απαιτήσει στους παραγωγούς τρίτων χωρών ή μόνο στους Ευρωπαίους και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς και καταναλωτές και να μην ε, δίνουμε καμία σημασία στην μη τήρηση των κανόνων από τρίτες χώρες. Τώρα το θέμα της γεωγραφικής προέλευσης. Θα πάψουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε χώρες ιδιαίτερα αναπτυγμένες όπως οι πολιτείες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κάποιες γεωγραφικές ενδείξεις ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ερνάντας Γκαρσία. Η παρέμβασή σου πραγματικά προκαλεί περαιτέρω συζητήσεις. Ο... Εμεί πάντα Ευρώπη είχαμε αυτές τις ανησυχίες, αυτούς τους φόβους να βλέπουμε τις νομές πολιτείες με τρόπο αυτοπεριοριστικό θα έλεγα κάτι το οποίο δεν έχουν πράξει οι ΗΠΑ. Ε, θα είμαι λοιπόν περίοδος να δω ποιες θα είναι η επιλογή που θα κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση για το Farm Bill όπου χορηγούσε για τη Γεωργία 77 δις δολάρια. Δεν είναι ποσό πολύ διαφορετικό από αυτό που χορηγεί η ΚΑΠ και υπενθυμίζουμε ότι εμεί έχουμε 10 εκατομμύρια γεωργών ενώ οι ΗΠΑ έχουν 2,2 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν βλέπετε η ενίσχυση ανά Γεωργών είναι πολύ υψηλότερη στις ΗΠΑ. Αυτό συχνά το ξεχνάμε. Θα πρέπει λοιπόν όμως να το υπογραμμίζουμε και θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή περίπτωση για Ερνάντα Γκαρσία. Άλμπερτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον, τον προηγούμενο μιλητή για την παρουσίαση της έκθεσης. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Γεωργία να βρεθούν λογικές λύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο παρά η υπογραφή δημερών συμφωνιών όπου συνήθως κάνουμε παραχωρήσεις. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν ε, οι κατάλληλες, ε, τα, τα, συνθήκες για να γίνουν σωστές διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ. Αυτό που, μου, που, με στεναχωρεί είναι ότι λείπουν τα πρότυπα μέσα στον ΠΟΕ. Δεν αρκεί στόχος του ΠΟΕ να είναι η διεύρυνση του εμπορίου, αυτό και μόνο. Θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα κριτήρια βάσει των οποίων να μπορούμε να μετρήσουμε. Τα πρότυπα που χρειάζονται για την προστασία καταναλωτών, περιβαλλοντικά πρότυπα, μαζί με τα εμπορικά πρότυπα, τα οποία λείπουν. Δεν είναι δυνατόν η Κομισιόν να δρά, να λαμβάνει μέτρα ε, κατά ενός Ευρωπαίου παραγωγού όταν έχει χαθεί ένα ε, ε, ενότιο από, ένα βόδι, έχει χάσει τη σήμανσή του δηλαδή και να τιμωρείται ο παραγωγός. Αυτό το οποίο πρέπει να απασχολεί την Κομισιόν είναι όλη η παραγωγή βοηδών και επίσης η εισαγωγή βοηδών από το εξωτερικό όταν σπάσονται τα ζώα έξω και εισάγονται τα κρέατα εδώ. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι εμείς θα δηλίζουμε τον κόνοπα όταν διεθνώς οι παραγωγοί μας μειονεκτούν και δέχονται διακριτική ε, μεταχείριση μέσα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Είναι λάθος να επικρίνει κανείς συνεχώς την Ευρώπη η έχω αναφέρει ε, τους αριθμούς. Η Ευρώπη απορροφά 90% των γεωργικών εξαγωγών της Αμερικής και 55% της, Νότια της ε, Νότιας Αμερικής. Ε, η, μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των βόρειο-αμερικανικών εξαγωγών έρχεται εδώ. Και εμείς μιλάμε τώρα για ελεύθερο εμπόριο για προσπαθήστε εσείς να εισάγετε λουκάνικα από τη Βαβαρία στην Αμερική, θα δείτε ε, ότι θα χτυπήσετε το κεφάλι σας στον τοίχο. Οι πόρτες θα είναι κλειστές. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτή την ε, κατάσταση. Και για να μην μακρηγορώ, αν θυμόσαστε τον Helmut Kohl, τον μεγάλο Ευρωπαίο και Γερμανό καγκελάριο, και να παραθέσω τι είχε πει σε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Γερμανία ε, σε πάνω από χίλιους ειδικού ε, του εμπορίου είχε πει ο Κόλ τότε εύχομαι να έχουμε τις ίδιες συνθήκες εισαγωγής τροφίμων στην Ευρώπη όπως υπάρχουν και για τις εισαγωγές αυτοκινήτων και επικράτησε απόλυτη υγεία στο κρατήριο διότι εννοούσε ο Κόλ ότι οι Αμερικανοί, οι Κορεάτες, οι Ιαπωνέζοι μπορούν να εισάγουν τα αυτοκίνητά τους μεν στη Γερμανία αλλά μπορούν να τα οδηγήσουν μόνο όταν τηρούν τις αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές. Το ίδιο θέλω και εγώ και για τα τρόφιμα. Να εισάγονται ξένα τρόφιμα μη ευρωπαϊκά στην Ευρώπη, αλλά να κυκλοφορούν και να διατίθενται μόνο όταν ανταποκρίνονται στις δικές μας προδιαγραφές. Εντάξει, να επιτρέπουμε ε, εισαγωγέ από την Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία ή τη Βραζιλία, αλλά μόνο εάν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Γι' αυτό επιμένω ότι στον ΠΟΕ πρέπει να υιοθετηθούν ξεκάθαρα πρότυπα στα οποία μπορούμε να συγκρίνουμε την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου που ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Εμείς δεν θέλουμε προστατευτισμό, επιθυμούμε οι κανόνες να είναι οι αυτοί. Διαφορετικά αυτό ονομάζεται στρέβλωση ανταγωνισμού. Ο Ζωζέ Μποβέ έχει το λόγο. Θα ήθελα να λάβω το λόγο στην συζήτηση. Ο συνάδελφός μου άνοιξε το δρόμο μιλώντας για λουκάνικα. Υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως μετά από την συμφωνία που υπήρξε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ΕΠΑ για τα βοηθεί με ορμόνες που δεν πρόκειται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς ε, ως ε, παραγωγή κρέατος ε, φορολογούμε θα με δασμούς 100% προτού να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Εμπιστούς αυτό είναι κρίμα θα έλεγα. Τώρα μιλάω επί της ουσίας. Τον Δεκέμβριο, Νοέμβριο, όταν θα διεξεχούν οι συζητήσεις στην Γενέβη, θα έχουν συμπληρωθεί 10 χρόνια μέρα με τη μέρα από την διεξαγωγή του διάσκεψης του Σιάτλ και τότε το 1989 το Δεκέμβρη είχαμε εξηγήσει πως ε, το ζήτημα των συμφωνιών επί του εμπορίου θα αντιμετώπιζαν πάντα το πρόβλημα της γεωργίας. Ε, θα το βρίσκαν μπροστά τους. Και εδώ και 10 χρόνια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το πρόβλημα της γεωργίας ε, επισκιάζει όλα τα άλλα ζητήματα για έναν λόγο το το όψη μου ότι η γεωργία δεν είναι ούτε αυτοκίνητα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε ψυγεία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί το ζήτημα της γεωργίας και να επιληθεί όπως επιλύεται πρόβλημα των βιομηχανιών. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι σημαντικό το μάλλον ε, διότι υπάρχει 8%, της, 8 της παραγωγής, 8% της παραγωγής που κυκλοφορεί από Ήπειρο σε Ήπειρο. Μειώθηκε. Προετών ήταν 10% αυτό το ποσοστό, τώρα είναι 8% και εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Ευρώπης αλλά με το σύνολο των εταίρων μας. Γιατί λοιπόν σήμερα επιβάλλουμε στις χώρες να αλλάξουν τη γεωργική τους πολιτική για 8% της παραγωγής η πραγματικότητα της παραγωγής στην Ευρώπη είναι ότι εμείς έχουμε τη γεωργία για να θρέψουμε τους πληθυσμούς μας. Το θέσμα των εξαγωγών είναι μια άλλη λογική. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν τους κανόνες της αγροτικής πολιτικής μόνο και μόνο έχοντας κατά νου τις εξαγωγές. Αυτό όμως γίνεται σε διεθνές επίπεδο για το 8% και όλοι οι κανόνες της ε, του ΠΟΕ για την ΚΑΠ οδήγησαν σε μια αλλαγή των κανόνων για το 8%. Το 92, ε, το 99, το 2003 και τώρα ξεκινάμε για μια νέα μεταρρύθμιση για να προσαρμοστούμε σε ένα άνοιγμα των αγορών που είναι μια υποθετική, ένα υποθετικό άνοιγμα που δεν τα αποκρίνεται στην πραγματικότητα της ε, αγοράς γεωρικών προϊόντων και της ε, αγροτικής κατανάλωσης. Θεωρώ λοιπόν πως εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα σε βάθος του προτού να επανελθούν οι συζητήσεις τον Δεκέμβριο. Όπως επίσης και με το όργανο <clears throat> επίλυσης διαφορών εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο είναι ένα κάκιστο εργαλείο, διότι οι επιλύσεις διαφορών, οι κυρώσεις περιπτώσει διαφορών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν παρά μόνο ανάμεσα σε πλούσιες χώρες. Εάν μια φτωχιά χώρα, φτωχή χώρα ε, κερδίσει απέναντι στις ΗΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να, ε, να λάβει οι κυρώσεις και με αυτό δεν θα έχουμε προβλέψει πως ακόμα και σε σε διαφορές και οι μικρές χώρες μπορούν να κερδίσουν, θα έχουμε ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει τη δικαιοσύνη και την ισότητα ανάμεσα στα κράτη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω πως τον Δεκέμβριο δεν θα επιτευχθεί συμφωνία, διότι ορισμένα κράτη, ειδικά... venire Luis. Luis Cabra Αναμφίβολα αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, οπότε πρέπει να γίνει εις βάθος συζήτηση. Νομίζω όμως ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν είναι η σωστή ώρα ούτε και το σωστό μέρος για να κάνουμε μια τέτοια ενδελεχή συζήτηση. Αλλά χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία γίνεται για να έχουμε για να έχουμε εφόδια και να κάνουμε αυτήν την συζήτηση που χρειαζόμαστε. Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλη την παρουσίαση. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά στοιχεία που μου φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι, πρέπει να κάνει τώρα που θα αναλάβει τις εξουσίες της συναπόφασης. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να ανταπεξέλθουμε στις τωρινές προκλήσεις ε, και υπάρχουν αιτήματα σε ε, τοπικό και σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να απαντήσουμε και στα δύο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια στρατηγική ούτως ώστε να αναπτύξουμε την τοπική παραγωγή με ό,τι αυτό ε, συνεπάγεται για την καταπολέμηση και των κλιματικών αλλαγών κτλ. Ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσουμε το ε, διεθνές εμπόριο που θα είναι ρυθμισμένο όπως επιθυμούμε. Ε, εάν υπάρξουν ελλείψεις, αν δεν υπάρξουν επαρκείς κανόνες στο διεθνές εμπόριο, θα είναι πάρα πολύ αρνητικές οι επιπτώσεις. Έχουν γίνει διαδοχικές μεταρρυθμίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει ακριβώς αυτό το μήνυμα τώρα. Θα δούμε ε, αν ε, η νέα κυβέρνηση στη ΣΥΠΑ θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας. Έχουμε δει κάποια θετικά μηνύματα βλέποντας και την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και θεωρούμε ότι με αυτά τα μηνύματα οδεύουμε, φαίνεται να οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και συμφωνώ με τη συνάδελφο που τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να εισαγάγουμε και την κοινωνική συνιστόσα ε, στα κριτήρια κατανομής ε, των ενισχύσεων. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να τοποθετηθεί η συζήτηση της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής. Καλωσορίζουμε αυτή την πρόταση. Εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε για αυτή και ελπίζουμε να συμβάλλει το ώστε η ευρωπαϊκή πολιτική να δώσει μια συνολική απάντηση για αυτήν την απαιτούμενη συμφωνία για να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση. Ελπίζω όλοι οι παγκόσμιοι φορείς να σταθούν σε θέση να λάβουν υπόψη το τωρινό πλαίσιο και να καταφέρουν να καταλήξουν σε αυτή την συμφωνία που είναι απαραίτητη δεδομένη κατάστασης. Grazie Luis, chiude la serie di interventi. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μαγκίνες και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο ΠΟΕ δεν έχει δεν απουσιάζει από τις συζητήσεις. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που μιλούν για τα ζητήματα της παραγωγής, ε, κάτι το οποίο δεν συζητιέται ακόμα στον ΠΟΕ και έχουμε κάποιο πρόβλημα να πείσουμε τους παραγωγούς μας ε, ότι θα πρέπει να κάνουν θυσίες. Η παραγωγή όπως και η παραγωγή γαλακτικών προϊόντων που συζητάμε σήμερα το πρωί έχουν ε, προβλήματα, είναι πολύ δύσκολο να τους πείσουμε για περαιτέρω θυσίες. Από ό,τι ακούσαμε υπήρξαν κάποιες ε, θετικές ε, επιπτώσεις, αλλά ακούσαμε επίσης ότι δεν μπορούν να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του γύρου της Ντόχα για τα προϊόντα. Με ανησυχεί επίσης ότι μαζί με αυτές τις ε, συζητήσεις ε, συζητάμε και το θέμα της μεταρρύθμισης ε, της κοινής αγροτικής πολιτικής, τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό. Υπάρχουν και οι προτάσεις του Φρανς για καλύτερη ρύθμιση των αγορών και των τιμών, κάτι το οποίο δεν συνέβη όμως στην Γεωργία και θα πρέπει να σκεφτούμε ιδιαίτερα το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη διότι συνεχίζουμε να διαβάζουμε και να ακούμε ότι χρειάζεται περισσότερη, περισσότερα γεωργικά προϊόντα, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει δυνατότητα επιβίωση των γεωργών μας. Έχω την εντύπωση πως η Κομισιόν θέλει να κάνει το καλό παιδί, το μαθητή της τάξης, υποβάλλει προτάσεις ε, αλτρουιστικού χαρακτήρα πολλές φορές και ξεχνάει εμάς τους ίδιους, την Ευρώπη δηλαδή. ανοίγει όλα τα χαρτιά και φτάνουμε στις διαπραγματεύσεις με όλα τα χαρτιά μας ανοιχτά. Αυτό δεν είναι σωστή διαπραγμάτευση. Θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνουμε σε μια συμφωνία που θα δεν θα αποβεί εις βάρος της γεωργικής παραγωγής. Αυτό ανησυχεί τόσο εμάς αλλά και ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ Μαγκίνης. Και τώρα ο κύριος Ταριό, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να εξετάσουμε τη μελέτη. Δεν... Μόλις τη λάβαμε, οπότε προς το παρόν δεν θα κάνουμε ούτε καν προκατακτικά σχόλια. Πρόκειται για μια τολμηρή απόπειρα για να γίνει μια γενική επισκόπηση του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσει. Θα το εξετάσουμε το κείμενο εντελεχώ και θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια στο μέλλον. Δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Ευχαριστούμε του συντάκτε τη μελέτη, ε, όλου του ε, παρεμβαίνοντε συναδέλφου. Ε, Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν ε, αποτελεσματική για να ξεκαθαρίσουμε τις ιδέες μας και τώρα που έπρεπε στο σημείο 7 της μεστής διατάξεως εισαγωγές βοήου κρέατος ε, προερχόμενε από τη Βραζιλία. Δεν πάμε και πολύ μακριά δηλαδή, πάντα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ε, πρόκειται για ένα αίτημα του κυρίου Γκαρσία. Έχει κληθεί ένα εκπρόσωπο ε, της υπηρεσία του Δουβλίνου για τα τρόφιμα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, ο οποίος θα μα αναφέρει σχετικά με το θέμα της αγωγής βοηού κρέατος στη Βραζιλία. Καλωσορίζω τους ε, εκπροσώπους τόσο του υπηρεσίας του Δουβλίνου όσο και τη Κομισιόν. για, που θα μας μιλήσουν για το σύστημα ελέγχου στην Βραζιλία αλλά και το σύστημα πιστοποίησης για την εξαγωγή κρέατος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά, όπω καταλαβαίνετε, εντάσσονται και στο πλαίσιο τη συζήτηση που είχαμε προηγούμενα, αναφορικά με την τήρηση των κανόνων. Να υπενθυμίσω στα νέα μέλη, τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με αυτού του συζητήσει, πω πέρυσι είχε υπάρξει με αποκλεισμό της εισαγωγής κρέατος από τη Βραζιλία σύμφωνα με κάποια αισθήματα που άπτονται της ε, ειχνηλασιμότητας και της πιστοποίησης. Οι περιορισμοί λοιπόν ε, των εισαγωγών περιορίστηκαν κατά τη και σε ορισμένες ε, εγκαταστάσεις μετά από τους ελέγχους που έγιναν από την αρμόδια υπηρεσία, κτηνοτροφική υπηρεσία του Δουβλίνου, αλλά ακόμα βρισκόμαστε σε, σε κάποιο πλαίσιο περιοριστικό. Έγιναν λοιπόν κάποιες απαλλαγές. Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, ευαίσθητο πάρε σε σχέση με την τήρηση των κανόνων που προαναφέραμε και θα χρειάζεται να εξεταστούν και να αξιολογηθούν από κοινού. Θα δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στους εκπροσώπους της Κομισιόν, ο κύριος από το και ο κύριος ε, Γκέτεμ από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα την κατάσταση της Βραζιλίας και την πολιτική που έχουμε στις εισαγωγές βοήου κρέατος από τη Βραζιλία. Η κοινότητα έχει μια πολύ αυστηρή ε, πολιτική εισαγωγών για τέτοιο κρέας και τα πιο αυστηρά μέτρα αφορούν την, ε, τον, αυθόδη, τον αυθόδη πυρετό. Θα θυμόσαστε ε, ότι είχε ξεσπάσει η ασθένεια αυτή και παρακολουθούμε με πολύ προσοχή ε, τυχόν ε, κρούσματα αυθόδους πυρετούς. Και ε, πυρετού. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύουμε τις εισαγωγές όταν έχει παρουσιαστεί κρούσμα για ένα έτος. Και εισάγουμε κρέας από περιοχές που δεν έχουν αυθέδει πυρετό Αμερική και Καναδά, Βόρεια Αμερική, ΙΠΑ δηλαδή και Καναδά, ε, Νότια Αμερική, ε, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Βραζιλία. Από την Αφρική κάνουμε εισαγωγέ βοήου από την Ναμίβια, Μποτσουάνα και ε, Νότια Αφρική και βεβαίως από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι οι μόνες χώρες από όπου επιτρέπουμε εισαγωγέ βοήου κρέατος, επειδή ακριβώ έχουμε επιβάλει αυτά τα απαγορευτικά μέτρα σε περιπτώσεις αυθόδου πυρετού. Έχουμε επίσης ε, πολύ ε, αυστηρά μέτρα όσον αφορά τα ε, υπολείμματα, ε, ε, ε, κτηνιατρικών φαρμάκων, μέτρα τα οποία στοχεύουν στην εξασφάλιση ότι τα κρέατα αυτά δεν έχουν υπολείμματα απογορευμένων ουσιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, έχει επίσης μία δέσμη πολύ αυστηρών μέτρων, τα οποία λαμβάνουμε επίσης υπόψη το κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες στην κοινότητα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν υπογραφεί από έναν επίσημο ε, κτηνίατρο ε, και υφίστανται ελέγχου στα σύνορα. Έχουμε λοιπόν το κανονικό καθεστώς ελέγχων ε, προϊόντων ε, ε, στα σύνορα για το κρέας το οποίο θα εισαχθεί στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, για να προλάβουμε τυχόν προβλήματα και για την ενίσχυση των, της ποιότητας ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ζώα δεν διατρέφονται με άλλα ζωικά προϊόντα και τυχόν ζωικά υπολείμματα δεν θα δοθούν ως ζωοτροφές ε, στα ζώα. Ε, θα θυμόσαστε και την, τις μεγάλες ε, οι επιδημίες ε, ε, γρήπης των χείρων που είχε εμφανιστεί στη Γερμανία λόγω της επειδή δόθηκαν ζωικές ζωοτροφές στα ζώα. Για να επανέλθουμε τώρα στη Βραζιλία. Όπως είπε ο πρόεδρος, στην αρχή του 2008 και μετά από διάφορους ελέγχους που κάνουμε στη Βραζιλία η Κομισιόν αποφάσισε να επιβάλλει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα, αυστηρές προδιαγραφές στις εξαγωγές βοήου κρέατος από τη Βραζιλία. Ποια είναι αυτές οι προδιαγραφές. Πρώτον, το κρέας θα πρέπει να είναι ε, σιτεμένο και χωρίς κόκαλα. Γιατί διότι εάν υπάρχει κάποιος ιός αυτόδου σπύρετου θα ε, εξουδετερωθεί με αυτόν τον τρόπο. Κοιτά, ε, βλέποντας τώρα τις ε, προτάσεις του ΠΟΗ και τους συναφείς κανονισμούς για την εμπορία και εισαγωγές κρέατων, το κρέας χωρίς κόκαλα και το σιτεμένο κρέας μπορεί να εισαχθεί ακόμα και από χώρε όπου υπάρχει αυτό ο δυσπύρετο. Εμείς έχουμε διάφορα επίπεδα, πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας και οι περιοχές της Βραζιλίας από, την οποία, από τις οποίες εισάγουμε βόλιο κρέας δεν έχουν αυτό, κρούσματα αυτόδους εδώ και ένα χρόνο, πέραν του ενός έτους. Πέραν αυτού όμως ζητούμε να είναι το κρέας ε, χωρίς κόκαλα και σιτεμένο. Τα ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση και πηγαίνουν στο σφαγείο, άλλα πρόσθετα μέτρα, θα πρέπει να κρατηθούν, να μείνουν τις τελευταίες 40 μέρες στην εκμετάλλευση εκτροφής και θα πρέπει να έχουν μείνει στην περιφέρεια, δηλαδή όχι στην εκμετάλλευση, αλλά στην περιφέρεια αυτή που είναι ελεύθερη τους πυρετούς, για τρεις μήνες. Λοιπόν, τρει μήνες στην περιφέρεια, χωρίς αυθόδη πυρετό και 40 μέρες πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση. Εκτροφής. Ε, για να εξασφαλίσουμε τώρα ότι αυτές οι 90 μέρες και 40 μέρες γίνονται σεβαστές και ότι συμμορφώνονται ή ε, εκτροφή στη παραγωγή, χρειάζεται ένα σύστημα ανείχνευσης. Και οι επιθεωρητές μας υιοθέτησαν ένα τέτοιο σύστημα στο τέλος του 2007 και στις αρχές του 2008 υιοθετήσαμε περαιτέρω μέτρα για την εισαγωγή βοή από τη Βραζιλία. Ποια είναι αυτά τα περαιτέρω επιπρόσθετα μέτρα εκτός από τους κανόνες των 90 και 40 ημερών. Πέραν αυτών λοιπόν είπαμε ότι όλα τα ζώα πρέπει να προέρχονται από ταυτοποιημένες ειδικέ μονάδες οι οποίες έχουν την σφραγίδα έγκριση των γενομικών υπηρεσιών έτσι ώστε να είναι όλες οι, εκτροφι... οι μονάδες εκτροφής καταχωρημένες στο σχετικό αρχείο και ε, να μπορούμε λοιπόν εύκολα να και γρήγορα να ταυτοποιούμε τα ζώα. Πριν ε, λοιπόν από την εφαρμογή αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων, πριν από το 2008, υπήρχαν πάνω από 30.000 ε, εκμεταλλεύσεις που είχαν περιληφθεί στο αρχείο αυτό και οι οποίες μονάδες ε, είχαν την άδεια εξαγωγής. Από τη στιγμή λοιπόν που εφαρμόστηκαν και τα πρόσθετα μέτρα στη Βραζιλία, από τις 30.000 μονάδες παραμείναν μόνο 100 μετά από τους ε, ελέγχους των ε, επιθεωρητών της Βραζιλίας. 100 λοιπόν ομάδες που είχαν άδεια εξαγωγής. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε το 2007 με το 2008, θα δείτε ότι το 2007 είχαμε περίπου 300.000 τόνους ε, κρέατος που εξήχθη από τη Βραζιλία στην κοινότητα, ενώ μετά από τις ε, ρήτρες ασφαλείες είχαμε λιγότερο από 10.000 τόνους το χρόνο. Δραστική λοιπόν μείωση των ποσοτήτων εξαγωγής βοήου κρέατος από τη Βραζιλία. Σας είπα λοιπόν για, τα 100, για τις 100 αυτές μονάδες που έμειναν στο αρχείο, στον κατάλογο και πριν, πριν ονομαστούν αυτές οι 100 μονάδες Ζητήσαμε ε, οι, οι βραζιλιανικές ε, αρχές να μας ε, παρουσιάσουν τις διαδικασίες ελέγχου τις οποίες εφαρμόζουν. Κάποιο... Αυτή η ρήτρα ασφαλείας λοιπόν έχει εφαρμοστεί πάνω εδώ και 18 μήνες και αυτή τη στιγμή στα αρχεία βρίσκονται 1.300, εκμεταλλεύσει εκμεταλλεύσεις από τις οποίες τα ζώα μπορούν να πάνε στο σφαγείο και, για να εξαχθεί το κρέας τους. Ε, αν δείτε τώρα το μέγεθο της Βραζιλίας και ε, την, μετά από την αποστολή της, ε, που, που έγινε των ε, στελεχών μας στη Βραζιλία ε, τα 1.300-1.300 μονάδες, εξαγωγικές μονάδες δεν είναι πολλές σε σχέση με τα μεγέθη της Βραζιλίας. Ο επιθεωρητής μας λοιπόν που επισκέφθηκε επιτόπου της μονάδες το 2008 πάνω από 8 φορές γιατί είχαμε πάνω από 8 αποστολές στη Βραζιλία, όχι μόνο τους ελέγχους του κρέατος, αλλά και για άλλα προϊόντα. Και η Βραζιλία σίγουρα είναι η χώρα την οποία έχουν επισκεφθεί τις περισσότερες φορές οι επιθεωρητές μας. Οι έλεγχοι που έγιναν πέρσι δεν αποκάλυψαν καμία ανησυχητική κατάσταση και δεν έτσι δεν ζητήθηκε, δεν είχε ε, λόγο η Κομισιόν να επιβάλλει άλλα συμπληρωματικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, βάσει ε, της αποστολής του Σώματος Επιθεωρητών που εδρεύουν στην Ιρλανδία και βάσει των συμπερισμάτων του FVO που έγινε, ε, μετά από τις επισκέψεις αυτές δεν χρειάστηκε η υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων. Η Κομισιόν βέβαια θα διατηρήσει την πολύ στενή παρακολούθηση το, της αγωγής των προϊόντων αυτών από τη Βραζιλία για να εξασφαλίσουμε ότι η δημόσια υγεία εξασφαλίζεται και η υγεία των ζώων βεβαίως και ότι υπάρχει πλήρης προστασία και των δύο πλευρών. αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, σας έκανα μια συνολική ανασκόπηση του τομέα και τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Κυρία Εράνς Sí, pues muchas gracias, señor Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο τι σημαίνει αυτή η προσεκτική επιλεκτική προσέγγιση της Κομισιόν. Τώρα, μετά από τη μελέτη που έγινε φέτος ε, από την υπηρεσία, την κτηνιατρική, διαπιστώνεται ότι το 50% των εκμεταλλεύσεων που ελέγχθηκαν στην Βραζιλία παρουσιάζουν παρατυπίες ε, Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε λοιπόν σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις προβλήματα σχετικά με την ίχνη δασιμότητα και για την χρησιμοποίηση του αυτού ατόμου σε διάφορες θέσεις, δηλαδή και του κτηνοτρόφου και του, ε, ε, ε και του ελεκτή αλλά και του ελεγχόμενου. αυτό δεν ε, μπορεί να συμβαίνει. Το θέμα της ε, πρόθεσης ε, κάποιων προϊόντων σε τρίτες χώρες μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης που συχνά δεν έχουν και τα κατάλληλα πιστοποιητικά και βρίσκονται από περιοχές που όπως αναγνώρισε και ο υπάλληλο τη Κομισιόν δεν είναι περιοχέ από τι οποίε επιτρέπεται η, είσοδος, η εισαγωγή κρέατο στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι αυτέ οι εξαγωγέ δεν είναι διόλου ελεγμένε και νόμιμε, διότι είναι κρέατο που έρχεται από περιοχέ οι οποίε δεν έχουν ελεγχθεί. Το θέμα τώρα της, του αυθόδους ε, πυρετού είναι ένας κίνδυνος ο οποίος μπορεί και να μας ε, πλήξει με, σύμφωνα με το κρέας το οποίο εισαγάγεται. Γι' αυτό συμβαίνει για το, στο 50% των εκμεταλλεύσεων και αυτό είναι επαρκής λόγος για να αναρωτηθούμε αν οι υπόλοιπε εκμεταλλεύσεις που δεν ελέγχονται πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξαγάγει προς την Ευρώπη. Πέραν των αποτελεσμάτων αυτών, σας δηλώνω ότι 50% των ελεγμένων εκμεταλλεύσεων παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Εν ώψη λοιπόν αυτού του αποτελέσματος δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό για τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους να τους απαιτούμε τέτοιες συνθήκες οι οποίες όμως δεν πληρούν από τις τρίτες χώρες και να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μετά από τόσες ελλείψεις και παρατυπίες δεν θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόσουν περιορισμούς στις εξαγωγές Βραζιλίας. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρεί τις υποχρεώσεις της για προστασία του καταναλωτή από τόσο προφανείς κινδύνους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σμίθ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους από την Επιτροπή για την παρουσίαση. Θυμάστε από την προηγούμενη θητεία ότι είναι ολόκληρη τελενοβέλα το θέμα του Βοή από την Βραζιλία και είχαμε δει διάφορα επεισόδια και νομίζαμε ότι όλα πηγαίνανε καλά και ξαφνικά επιβάλλεται πλήρη απαγόρευση ε, των εισαγωγών. Χαίρομαι λοιπόν που ακούμε την παρουσίαση γιατί ε, εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση, η εκτροφή μας το ίδιο και εσείς παρακολουθείτε τη Βραζιλία τι κάνει. Αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα του κρέατος και την ανοιχτή ανιχνευσιμότητα. εύλογε ανησυχίες υπάρχουν, όπω είπε και η κυρία Γκαρσία, κρεμούν σοβαρά ζητήματα στον τομέα αυτό και δεν θέλουμε επανάληψη των ίδιων επεισοδίων. Έχουμε περάσει από τις 30.000 στις 1.300 καταγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις και έχουμε περάσει 10.000 τόνους κρέατος ε, δηλαδή δεν είναι και τόσο σημαντικό το ζήτημα όπως το παρελθόν. Αλλά αν ακόμη ε, ε, υπάρχουν ερωτηματικά για την ποιότητα και λέτε ότι στο 50% των επιθεωρήσεων δεν περνάνε το τεστ, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Καλά κάνουμε και παρακολουθούμε τι γίνεται στις επιθεωρήσεις σας, γιατί έτσι μπορούμε να σας θέτουμε και ερωτήματα. Άλλο ε, παρατυπή, άλλο να μιλάμε για παρατυπίες και άλλο να μιλάμε ε, για κάποια παράληψη. Τι έλειπε, ένα χαρτάκι ή ένα έντυπο ή υπήρχε σοβαρό πρόβλημα παρατυπίας, ε, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε, πρέπει να δούμε οι λέξεις που χρησιμοποιείτε σε τι αντιστοιχούν. Θα ήθελα να μας καθησυχάσετε. Γιατί και στην Ιρλανδία και στη Σκωτία οι εκτροφείς μας ανησυχούν ιδιαίτερως ε, για αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν είχαμε προβλήματα με τις εισαγωγές του βοηοκράτους από τη Βραζιλία, αρκεί να πληρούνται τα ίδια πρότυπα. Πρέπει οι εκτροφείς μας να ξέρουν ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα. Ε, και όλοι περιμένουν μια απάντηση σε, σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντεσί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα, είχα αναφερθεί στη Βραζιλία και στην προηγούμενη συζήτηση με τον ΠΟΕ. Αναγνωρίζω τις προσπάθειες της Κομισιόν κατόπιν πιέσεών μας τα τελευταία δύο χρόνια. Απλώς δεν θα ήθελα να αναφερθούμε μόνο στη Βραζιλία. Υπάρχουν χώρες που έχουν παρουσιάζουν μεγαλύτερα ή ίδια προβλήματα με τη Βραζιλία. Έχω και εγώ επισκεφθεί τη Βραζιλία και μεγάλα σφαγεία εκεί. Τα σφαγεία αυτά έχουν ε, από πλευράς διαδικασίας και υγιεινής ε, καθαρά ευρωπαϊκά πρότυπα και πολλά μάλιστα είναι και καλύτερα. Επίσης έχω εξετάσει το θέμα της μεταφοράς ζώων στη Βραζιλία Λοιπόν, ε, άμα θέλετε να ξέρετε τα, τα, τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Βραζιλία, ε, Είμαστε πάρα πολύ μεγαλόψυχοι όσον αφορά τις συνθήκες μεταφοράς, αλλά πάρα πολύ αυστηροί όταν αφορά άλλες χώρες. Λοιπόν, ε, Υπάρχει μεγάλο ε, έλλειμμα ε, όσον αφορά τις συνθήκες, ιδίως το θέμα της μεταφοράς των ζώων και γι' αυτό χαίρομαι που, η Κομισιόν εφαρμόζει αυστηρά μέτρα, αλλά και μεγαλύτερη αυστηρότητα ακόμα δεν βλάπτει. Όταν συγκρίνω την Ευρώπη με τη Βραζιλία και άλλες χώρες, ε, σημειώνω το εξής. Όταν στη, δική μου περιφέρεια ε, ένας ε, ε, γεωργός ξεριζώνει 50 μέτρα φράχτη, τον κοπανάνε με ένα πολύ γερό πρόστιμο στο κεφάλι. Ενώ στη Βραζιλία, εάν σημειώσουμε σε μία εκμετάλλευση ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές και η εκμετάλλευση αυτή έχει 150.000 ζώα, θα πρέπει να υπάρχει μία αντιστοιχία ποινών ή κυρώσεων. Επίσης στην ε, επαρχία του Ρεσίφε που υπάρχει το, το τεράστι, η τεράστια μονάδα πετρολίνα ε, έχει κάνει μία αφέμαξη, ε, έχει χρησιμοποιήσει τόσο πολύ νερό από τα ποτάμια του Ρεσίφε ώστε να έχει τελείως αποκοπή ο, η είσοδος του νερού από τον Ατλαντικό. Εάν λοιπόν κάνουμε σύγκριση το, του μεγεθών της Βραζιλίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η κακή εκμετάλλευση των ε, πλουτοπαραγωγικών πηγών θα ήταν σαν να είχαμε στερέψει το Δούναβι στη Βουδαπέστη και, και, και, στην Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, είναι δύσκολη η σύγκριση τέτοιων μεγεθών μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με το τελευταίο σχόλιο του κυρίου Ντέστ και στην Επιτροπή Περιβάλλοντας το πρωί μίλησαν για τον Αμαζόνια, τις κλιματικές αλλαγές και το γίνεται στο ΦΑΟ. Ε, πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ε, πώς θα χειριστούμε το θέμα της αλλαγής του κλίματος διεθνώς, όχι μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, συγκεκριμένα για την έκθεση αυτή της Βραζιλίας, ε, εάν θυμόσαστε είχαμε 30.000 εκμεταλλεύσεις, έτσι με, ε, βοηδή. Και τώρα έχουμε ε, 1.300 εκμεταλλεύσεις. Βλέπετε λοιπόν την τεράστια μείωση μετά από τους ελέγχους και τους κανόνες της Κομισιόν. Ε, κατόπιν πολλών πίεσεων βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και των ελέγχων. Έξι ε, από τις μονάδες δεν είχαν συμμορφωθεί τρεις είχαν ε, παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την ταυτοποίηση των ζώων και πραγματικά εάν ένας Ευρωπαίος παραγωγός τον είχαν πιάσει με τέτοιες παραβάσεις θα του είχαν κλείσει την εκμετάλλευση. Εάν θέλουμε να τα πρότυπά μας να εφαρμόζονται 100% τότε πρέπει να έχουμε 1000% ασφάλεια στην ποιότητα των εισαγωγών. Δεν είμαι λοιπόν απόλυτα βέβαιη ότι τα συμπεράσματα της Κομισιόν είναι όλα πάνε καλά με λιγάλα η κατάσταση με τη Βραζιλία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω λεπτομέρειες των ελέγχων το επίπεδο των ελέγχων που γίνεται, δεδομένου ότι η Βραζιλία είναι μια τεράστια χώρα. Εγώ όταν είχα πάει είχα δει πάρα πολλά ε, ε, ζώα χωρίς ενότια ε, και ε, υπάρχουν ακόμα σαφώς ε, ζώα τα οποία δεν είναι ταυτοποιημένα. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο λεπτομερείς αναφορές. Ίσως να μην έχω διαβάσει καλά και τον, την έκθεση, αλλά έχω ακόμα σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των συναρμοδίων αρχών. Όταν ακούμε για αρμόδιες αρχές ε, και βλέπουμε τις αρμόδιες αρχές της Βραζιλίας και τις ονομάζει η Κομισιόν, πόσο ε, αξιόπιστες είναι αυτές οι, Βραζιλία, οι αρχές της Βραζιλίας. Ευχαριστώ. Κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Έχω ένα πρόβλημα λόγω των όρων που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην έκθεση. Αναφέρεστε, Φερρυπίν, σε ίσονο σημασία ελλείψεις και σε μη σημαντικέ ε, παραλήψεις Οι ατέλειε. Με προβληματίζουν αυτοί οι όροι. Άκουσα την Κομισιόν το πρωί, άκουσα τον κύριο Ντάζ, ε, παρευρέθη στην προηγούμενη συζήτηση, άκουσα τα, τις απόψεις των μεν και των δε και κάτι που είναι ξεκάθαρο όταν μιλώ εγώ με εκτροφής είναι ότι θέλουν να ξέρουν πως δεν θέλουν να ξέρουμε ότι δεν είναι κατά των εισαγωγών απλά πρέπει να πληρούνται τα ίδια πρότυπα όπως αυτά με τα οποία συμμορφωνονται εκείνοι ε, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό δεν γίνονται πλέον αποδεκτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά από τους εκτροφείς μας. Αυτή η έκθεση ουσιαστικά επαναλαμβάνει προηγούμενες υποσχέσεις από τις βραζιλιάνικες αρχές, ε, αλλά ουδέποτε εκπλήρωσαν αυτές τις υποσχέσεις τους. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για την ανείχνευση των... Αυτό το σύστημα που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία είναι αξιόπιστο για την ε, ανιχνευσιμότητα των ζώων. Σε αυτό θέλουμε να μας απαντήσετε. Διαβάζω μέσα στην έκθεση ότι από 50% των εκμεταλλεύσεων δεν συμμορφούνται με τις απαιτήσει. Ε, οπότε ε, όταν οι οικονομικοί φορείς, οι εκτροφείς ε, δεν καταθέτουν εγκαίρως, ε, καταθέτουν ετεροχρονισμένα τα συνοδευτικά έγγραφα των ζώων και 7 μήνες μετά την παραλαβή. Συγγνώμη, αυτά τι σημαίνουν. θα τους είχαν μαντρώσει τους δικούς μας τους εκτροφείς αν είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν πρόκειται για ίσονο σημασίας παραλήψεις εδώ. Μπορώ να σας ε, απαριθμίσω όλες τις ε, ατέλειες. Παραδείγματος χάρη ε, των ενωτιών 14, με 14 μήνες καθυστέρηση παραδείγματος χάρη. Εσείς επιλέξατε με τα δικά σας κριτήρια κάποιες εκμεταλλεύσεις ε, και εντάξει, αν συμμετείχαν στην επιλογή ε, συμμετείχαν μάλλον στην επιλογή και οι βραζιλιάνικες αρχές. Επέλεξαν τις καλύτερες και από τις καλύτερες εμείς βρήκαμε παράτυπες τις 50%. Το 50% των εκμεταλλεύσεων, ε, μα οι υπόλοιπες τι είναι που είναι οι χειρότερες. Πρέπει να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καλό θα ήταν να τελειώσει αυτό η κομμωδία. Να, πάμε, να πηγαίνουμε συνέχεια στη Βραζιλία και να επιθεωρούμε εκμεταλλεύσει που ποτέ δεν πρόκειται να συμμορφωθούν με τα πρώτα. Οι δικοί μα οι εκτροφεί ξεκάθαρα λένε ότι πλέον δεν δεχόμαστε εισαγωγές προϊόντων που δεν παράγονται με τα ίδια πρότυπα. Και ξέρετε ότι δεν πρόκειται για ίσονο σημασία σε αδικήματα ε, που μπορούμε να παραβλέψουμε. Ε, θα έπρεπε λοιπόν, εφόσον έχουν έτσι τα πράγματα, να απαγορευτούν τελείω οι εισαγωγέ από την ε, Βραζιλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Νικολέσκου. Αγαπητοί συνάδελφοι, για πρώτη φορά λαμβάνω το λόγο ενώπιον σας. Σήμερα το πρωί γράφτηκα μεγάλη καθυστέρηση και θα ήθελα να πω ότι την προσεχή φορά που θα έχουμε καλεσμένο επίτροπο θα πρέπει να στήσει το λόγο προτού να ξεκινήσει να μιλάει. Τώρα συμφωνώ με, τις, με τα όσα ακούστηκαν σχετικά με τον χαρακτήρα, τον άδικο, τον άνισο χαρακτήρα που υπάρχει δεδομένων των, των επικρίσεων που ασκήθηκαν από την Κομισιόν. Δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν που σήμερα μπορούμε να να ανοίξουμε τις ε, εισαγωγές μας ε, από τη Βραζιλία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένα στο πλαίσιο της Κομισιόν ή για αυτής της αίθουσας ε, μπορεί να κρίνει όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει κανόνες σε δεμάτα περιβαλλοντικά κλπ. που θα έχουν ως στόχο μόνο την κύρωση των παραγωγών μας, των γεωργών μας, των κοινοτρόφων μας όλοι συμφωνούμε πως αυτό που προέχει είναι η προστασία των καταναλωτών, της κοινωνίας μας, του περιβάλλοντός μας. Αλλά θα πρέπει να μου εξηγήσει για ποιο λόγο, εάν αυτό είναι ο στόχος, δηλαδή η προστασία του καταναλωτή, οι κανόνες εφαρμόζονται στην Ευρώπη και όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν στην Ευρώπη τα προϊόντα τους. Αν έχουμε ένα σύστημα όπου δεν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες σε όλους όσοι επιθυμούν να πολλούν προϊόντα στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι κοροϊδεύουν τους καταναλωτές. Αφήνουμε να εννοηθεί ότι οι ρυθμίσει που φασίζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα ισχύουν για όλα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην αγορά μας, στις αγορές μας, ενώ υπάρχει μια τρομακτική στρέβλωση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά προϊόντα και τα εισαγόμενα. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε μια οικονομία στο πλαίσιο της ε, μετέθεσης ΚΑΠ με δίχως την εφαρμογή της αμοιβαιότητας σε ό,τι φορά την εφαρμογή των ρυθμίσεων. Διαφορετικά είναι σαν να πέφτουμε με το κεφάλι στον τοίχο. Τώρα ακούσαμε το πρωί πως ε, εάν ε, δεν δεχθούμε την παραπλή συμμόρφωση τότε κυρώνουμε τους ε, καταναλωτές αλλά όχι τους παραγωγούς. Είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο. Λοιπόν, <clears throat> συγκεκριμένα. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν οι προραλήσαντες και το επιχείρημα το οποίο λέει ότι πρόκειται για προστατευτισμό εάν σκιζόμαστε παρόμοια επιχειρήματα νομίζω ότι αυτό είναι εσφαλμένο διότι αυτά τα οποία συζητάμε αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, του καναλωτή, των πολιτών μας και αυτό είναι κάτι που αποτελεί την βάση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευχαριστώ κύριε Μπεσού, κύριε Άγνιου. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω τον κοινικό τόνο αυτών ορισμένων παρατηρήσεων. Θα ήθελε Κομισιόν όταν πάει την επόμενη φορά να ρίξει ένα νόμισμα στο πάτωμα, στο χάρτη της Βραζιλίας και να πει εκεί θα πάμε. Τυχαίο δηλαδή έλεγχο και όχι προειδοποιημένος. Όσον αφορά τώρα την, το, το, να μην ε, ταΐζονται τα ζώα με ζωικά υπολείμματα, ε, τι γίνεται με τα υπολείμματα οστών, ε, σε κονιορ, κονιορ, κονιορτοποιημένα υπολείμματα οστών, παραδείγματος χάρη στις ζωοτροφές. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επίτροπη για όλα αυτά τα ωραία που μας είπε. Όμως φαίνεται ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε περάσει ε, ε, έχει, πο, πολλές ώρες με τη συζήτηση αυτή για τη Βραζιλία και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι χρειαζόμαστε ορισμένε βελτιώσεις επιτέλους και ε, η Κομισιόν ομιλεί βεβαίως με μία φωνή αλλά αυτό έχει συμβεί επειδή εμείς έχουμε πιέσει πολύ την Κομισιόν τέλος πάντων να ξεκινήσει όλες αυτές οι διαδικασίες. Τώρα αν ένας παραγωγός με ρωτήσει τι γίνεται με την αποθήκευση, με την εισαγωγή του κράτους από τρίτες χώρες και αν υφίσταται τις ίδιες διαδικασίες όπως και απαιτήσει όπως το ευρωπαϊκό κρέας. Αν με ρωτήσει λοιπόν αυτό και εγώ διαβάσω την έκθεση εν συνεχεία, η απάντησή μου θα ήταν ναι, μεν, αλλά. Και αυτή η απάντηση, ναι μεν αλλά, δεν αλέσει καθόλου στους παραγωγούς. Θέλουν να ξέρουν ή ναι ή όχι. Δεν μπορούμε όμως να απαντήσουμε ξεκάθαρα ναι, διότι οι Ευρωπαϊκή υπάρχουν ακόμα ελλείψεις στην πολιτική αυτή. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα μετά από αυτή την έκθεση. Θα εξετάσουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης και θα πούμε ότι ναι, έχουμε σημειώσει πρόοδο, δεν είναι ιδανική η κατάσταση, αλλά ε, υπάρχει πρόοδος και ε, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στους ελέγχους κλπ. Ή θα πούμε ε, έχει οδός και μπορούμε να διευρύνουμε τον κατάλογο των εκμεταλλεύσεων. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα να ξέρω την Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εφησυχάσουμε στις δάφνες μας και να πούμε ότι ε, έχουμε, έχει τελειώσει το ζήτημα. Οι έλεγχοι πρέπει συνεχώς να εντείνονται γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη λύση των προβλημάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διά, διάβασα την έκθεση αυτή του ΦΑΟ και ιδιαίτερα τα σημεία για το κρέας της Βραζιλίας και τα συμπεράσματα λένε ότι η κατάσταση γενικά είναι ικανοποιητική. Τώρα, εγώ ως καθηγήτρια Εάν ε, ένας μαθητής ή μία μαθήτριά μου μου έδινε μια τέτοια έκθεση, δεν θα της έβαζα καλό βαθμό. Ε, πρέπει να πω ότι ε, ενώ πολλοί είναι ικανοποιημένοι με την έκθεση αυτή και εγώ είμαι ικανοποιημένη, εάν δείτε τον κατάλογο περιεχομένου, περιεχομένου της έκθεσης και τα συμπεράσματα, θα δείτε ότι υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μία ανισότητα. Πολλά τα περιεχόμενα, αλλά στα συμπεράσματα Need action. Υπάρχουν συνεχείς παρεμβολές λόγω των κινητών τηλεφώνων. Γι' αυτό αναγκάζομαι και διακόπτω. Λοιπόν, όπως είπε ένας από τους προηγούμενους ομιλητής, αυτή αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας, διότι συνεχώς παρουσιάζονται εκθέσεις από τη Βραζιλία. 50% ε, των εκμεταλλεύσεων εκεί διαπιστώθηκαν παρατυπίες και επειδή η χώρα είναι τόσο μεγάλη θα πρέπει ας πούμε να κάνουμε έναν έλεγχο τυχαίο, να ρίξουμε μια καρφίτσα και όπου πέσει εκεί να κάνουμε τον έλεγχο. Εγώ δεν νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ικανοποιητική όπως πολλά άλλα μέλη εδώ στην Επιτροπή. Ο κύριος Γκλάτφελντερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Άλμπερτ Ντες ότι δηλαδή στην Βραζιλία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων, την καλή μεταχείρισή τους κλπ. Το Κοινοβούλιο πριν από μερικούς μήνες ενέκρινε ένα ψήφισμα, ένα κανονισμό για το ε, θέμα των προϊόντων φώκιας και ζήτησε οι φώκες να μην φωνεύονται με τον τρόπο με τον οποίο φωνεύονται σε κάποιες περιοχές του κόσμου κάτι το οποίο θεωρούμε ανήθικο και βίαιο. Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη λάβει, μέτρα σύμφωνα με τα οποία πτυχές ε, της ε, καλής μεταχείρισης ε, των ζώων ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγωγές. Και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο. Στον ΠΟΕ ίσως ε, να μην κατορθώσαμε να λάβουμε μια εντολή προκειμένου να κάνουμε αναφορές σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων αλλά εν τόσο γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο που αφορά στις φώκες για την απαγόρευση εισαγωγής. Θα μπορούσε να αποτελέσει λοιπόν μια πολύ καλή νομική βάση για τις εισαγωγές ε, κρέατος από την Βραζιλία. Τα πρότυπα λοιπόν σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων που απαιτούμε από τους δικούς παραγωγούς θα μπορέσουμε να τα απαιτούμε και από τους ε, κτηνοτρόφους ε, οι οποίοι εξάγουν τα προϊόντα του στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Ευρωπή προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά τα ερωτήματα. να εξετάσω τα σημαντικότερα εξ αυτών πρώτα-πρώτα. Μιλάμε για την διαμετακόμιση κρέας το οποίο διαμετακομίζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πληρεί τις ίδιες προϋποθέσεις που, που απαιτούμε και στις εισαγωγές. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρξει καμία παρατυπία Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενη παρατυπία λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Επαναλαμβάνω, τα, το κρέας που διαμετακομίζεται μέσω της Ευρωπαϊκής δηλαδή ερχόμενο από τη ΣΥΠΑ και με προορισμό της, ε, τη Ρωσία, θα πρέπει να πληρεί τις ίδιες προϋποθέσεις ως αν το κρέας να είχε εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι φορά την ανιχνευσιμότητα, πολλοί βουλευτές το έδειξαν. Φυσικά στην Βραζιλία θα δούμε πολλές ε, αγελάδες ε, δίχως ενότια. Μόνο 1% των εκμεταλλεύσεων πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και μπορούμε να γνωρίζουμε πως ε, στις ε, ε, εγκαταστάσεις αυτές υπάρχει ανεχνευσιμότητα. Παραλαμβάνω, 1% του ζωικού κεφαλαίου καταγράφεται. Μα φυσικά και υπάρχουν πολλά βοηθοί χωρίς ενότια στη Βραζιλία. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι το κρέας που εξάγεται προς την Ευρώπη να συμφωνεί με τις υποχρεώσεις ότι έχουν παραμείνει 40 μέρες τα ζώα στην συγκεκριμένη, 90 μέρες στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα εντάξει δεν συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να πάρουμε μια καρφίτσα και να την πετάξουμε σε ένα, σε ένα, πάνω σε ένα χάρτη. Ναι, εντάξει. Αλλά επιστώσει δεν κάνουμε ακριβώς έτσι τις, ε, τους ελέγχους μας, αλλά φτάνουμε απρόπτα και ελέγχουμε τις ε, εκμεταλλεύσεις. Και όχι μόνο σε τρίτες χώρες, αλλά δύο γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την ανιχνεσιμότητα του ζωικού κεφαλαίου στα κράτη-μέλη. Τώρα, σχετικά με την έκθεση, είναι καλή ή κακή. ...150 εκθέσεις ετησίως παράγουμε. 150 εκθέσεις, 150 έλεγχοι γίνονται... Οι, μισές, ε, οι μισή έλεγχοι γίνουν στα κράτη-μέλη, οι άλλοι υπόλοιπε έλεγχοι στο τρίτες χώρες. Μπορείτε να πάτε στο ιστοσελίδα μας και να ελέγξετε αυτές τις εκθέσεις. Οι ελεγκτές μας είναι επαγγελματίες, οι καλύτεροι στον κόσμο θα έλεγα. Και ποιος είναι ο σκοπός ε, και το έργο ενός ε, ελεγχθεί είναι να εντοπίσει πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά περιέχονται στις εκθέσεις και ο παρακαθισμένος μου που είναι ένας από τους καλύτερους ελεγχθές είναι έτοιμος να απαντήσει σε κάθε σημείο της έκθεσης. Το θέμα της ε, διατροφής των ζώων με υπολείμματα. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το ανεχόμαστε και στο εξωτερικό. Μία από τις χειρότερες επιδημίες του 1997-1999 για τον αυτόδη πυρετό όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε να σφαγιάσει 11 εκατομμύρια ζώα ξεκίνησε με αυτή την ε, διατροφή μέσω υπολοιμάτων και η πανόλη των χείρων, με συγγνώμη, ο πυρητός των χείρων, η γρήπη των χείρων και αυτή ε, προέκυψε από την διατροφή ζώων μέσω υπολοιμάτων. Γι' αυτό και απαγορεύτηκε. Ε, μιλήσαμε μετά και για τα σφαγεία τα σφαγεία στη Βραζιλία ε, πληρούν τα ανώτατα πρότυπα και ελέγχονται από τους ελεγχτές μας αλλά είναι πολλές φορές ε, υψηλότερης ποιότητας ε, από αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψη του Κοινοβουλίου πέρυσι τουλάχιστον οι βουλευτές που επισκέφθηκαν πέρυσι την περιοχή μπορούν να διαβεώσουν πως ε, η ποιότητα των σφαγίων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στην έκθεση την οποία εξάλλου ανάγνωσαν ε, και κάποιοι από τους κύριους κύριους βουλευτές αναφέρθηκαν παρατηρήσεις σχετικά με τις 6 ε, από τις 12 εκμεταλλεύσεις. Σε τρεις βρήκαμε ίσονο σημασία προβλήματα και σε άλλες τρεις ε, εντοπίσαμε πιο σημαντικά προβλήματα. Μπορώ να δώσω το λόγο στον Αντρέ προκειμένου να σας μιλήσει αναλυτικότερα για αυτά τα προβλήματα. Διαφορετικά θα παραμείνουμε εδώ στις θέσεις μας και θα είμαστε στη κάθε βουλευτή προκειμένου να απαντήσουμε σε ερωτήσεις του. Ωραία, σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, έγινε μια εκτενή συζήτηση. Οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει στο προηγούμενο σημείο σχετικά με τον ΠΟΕ δείχνουν την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουμε ε, σε θέματα που αφορούν στο άνοιγμα των συνόρων μας ε, προϊόντα τα οποία δεν τηρούν ευρωπαϊκούς κανόνες ενώ οι κανόνες αυτές την χάνουν απόλυτης τήρησης από τους ντόπιου παραγωγούς και φυσικά προσέχουμε πάρα πολύ να μην διολυστήσουμε στο προστατευτισμό. Εάν δεν υπάρχουν περαιτέρω παρατηρήσει, νομίζω ότι μπορούμε στο σημείο αυτό να ολοκληρώσουμε την ε, σημερινή μας συνεδρίαση και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Παρακαλώ στις 10. Όχι, διακόψη. Το συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. 9 οι συντονιστές και στις 10 όλα τα μέλη της Επιτροπής σε αυτή την αίθουσα. Καλό σας βράδυ.